Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο ε, γυναίκες συναδέλφους βλέπω αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όλους. Ας ε, συνεχίσουμε με την συνεδρία της Επιτροπής. Και ας πάμε στο σημείο 14 σύσταση για σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίνει την άνοιξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη σύμβαση για τη δημιουργία πολυμερού δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών. Το βήμα αυτό είναι σημαντικό. Προς, υπέρ του απόλυτου συμφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αφορά συζητήσεις ε, για τη συμφωνία ενδεχομένως στο πλαίσιο της TTIP με τις ΗΠΑ αλλά και στη συμφωνία με τον Καναδά. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλαμε να πάμε πιο πέρα από το σώμα ISDS ε, για την επίλυση των διαφορών το οποίο δεν χρησιμοποιούμε πλέον σε εμπορικές συμφωνίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταφέραμε να Καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το κομμάτι. Ήταν μεγάλη επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμάμαι πολύ καλά τις αρχικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου ο Επίτροπος ήταν αδύνατο να πιστεί ότι το ISDS ε, ανήκε στην ιστορία, στο παρελθόν. Κινήθηκαν όμως τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι συνθήκε πλέον τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στα κράτη-μέλη. Συνεπώ σήμερα ε, γίνεται συζήτηση για μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών. Θα περάσουμε από ένα διμερές σε ένα πολυμερές διεθνές σύστημα. Στη συμφωνία ΣΥΤΑ με τον Καναδά ε, έχουμε ένα κείμενο που καθορίζει ότι οι εταίροι θα προσπαθήσουν να καθιερώσουν, να δημιουργήσουν ένα πολυμερές δικαστήριο και αυτό αποτελεί το προϊόν συζητήσεων εδώ στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι μας οι εταίροι το έχουμε σημειώσει. Εγώ υπήρξα, ήμουν παρόν όταν, ε, όταν έγινε η παρουσίαση ε, σε μια διάσκεψη στο Ναϊρόμπι για ένα πολυμερές δικαστήριο. Στη συνέχεια ακολούθησαν ε, πολλές συναντήσεις προγνωμόνων. όπως φαίνεται αρχίζει να διαμορφώνεται ένα σύστημα προς αντικατάσταση του ISDS, ένα σύστημα ιδιωτικού δικαίου. Και για πολλές συμφωνίες ε, με πολλές χώρες αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τα εμπρός. Δεν ισχυρίζομαι ότι η εντολή που θα συζητήσουμε θα είναι το τελικό νομοσχέδιο, αλλά πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης, ε, θα μας το παρουσιάσει ο κύριος Κόλιν Μπράουν. Έχετε το λόγο κύριε Μπράουν, παρακαλώ. Um, um, Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για το Πολυμερές ε, Επενδυτικό Δικαστήριο. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να χωρίσω την παρουσίασή μου σε τρία μέρη. Πρώτα απ' όλα να σας κάνω μια σύντομη περιγραφή του πώς βλέπουμε εμείς ε, την ιδέα του ε, πολυμερούς δικαστηρίου. Αυτό σχετίζεται και με τα σχέδια οδηγιών ε, που εξετάζετε εσείς. Δεύτερον, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις εσωτερικές εξελίξεις. Τι έχουμε κάνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιο αυτό και τρίτον θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει εξωτερικά τι έχουμε καταφέρει να κάνουμε στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και με τις τρίτες χώρες. Για το πρώτο, στο οποίο ήθελα να αναφερθώ, ε, ποιο είναι το σκεπτικό μας η βασική δομή ε, την οποία έχουμε θέσει ως στόχος προέρχεται από την προσέγγιση που αναπτυχθήκε στο πλαίσιο της TTIP και που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της ΣΥΤΑ του Βιετνάμ και των λοιπόν διαπραγματεύσεων. Σκοπός λοιπόν είναι να συσταθεί ένα δικαστήριο το οποίο θα ε, ε, λειτουργεί ε, πρωτοβάθμια πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις λεπτομέρειες της κάθε υπόθεσης και δευτεροβάθμια σε με ένα σώμα για εφέσεις, για προσφυγές επιζητημάτων νομικών και λαθών επιγεγονότων και ε, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα των ε, αποφάσεων. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο μηχανισμό μέσα στον χρόνο θα βοηθήσει στη δημιουργία συνοχή και ε, προβλεψιμότητα. Τα δύο αυτά επίπεδα πιστεύουμε θα στελεχώνονται από δικαστέ πλήρου απασχόληση. Δηλαδή δεν θα έχουν καμία άλλη απασχόληση τα εν λόγω άτομα πέραν του να είναι δικαστές για το δικαστήριο αυτό για το επενδυτικό δικαστήριο και επίσης προβλέπουμε και κάτι άλλο ότι ότι θα είναι εμπειρογνώμονες σε ε, διεθνές δημοσιοδίκαιο και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί από τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στο σύστημα γνωρίζουν και έχουν εμπειρία ε, στο εμπορικό δίκαιο, στην εμπορική διαιτησία και εμεί πιστεύουμε ότι απαιτείται εμπειρία σε δημόσιο διεθνές, σε διεθνές δημόσιο δίκαιο, κάτι καταλληλότερο για να μπορέσει κανείς να εξισορροπήσει τα δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, όπως ε, είναι η περίπτωση ε, στις υποθέσεις αυτές. Ε, το βλέπουμε ακριβώς όπως το περιγράψατε, ως μια απομάκρυνση από αυτό που θεωρείται ιδιωτική δικαιοσύνη, αντόκ διαιτησία ε, μέσω εμπορικών μηχανισμών προς ένα μάλλον δημόσιο σύστημα. Ένα δημόσιο σύστημα το οποίο ε, θα βασίζεται στις δικές μας δικαστικές νομικές παραδόσεις και στις ε, παραδόσει που προωθούν σε άλλα διεθνή δικαστήρια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει και κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό ότι το σκεπτικό είναι να μην δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για ISDS. Έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι θα λειτουργεί με μια προσέγγιση ε, opt-in ε, προαιρετικής επιλογής. Έτσι λοιπόν αυτό το πολυμερές δικαστήριο θα ισχύσει για τις υπάρχουσες 2.300 ε, επενδυτικές συμφωνίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και πολύ μεγάλο το πεδίο εφαρμογή του, οπότε είναι σαφώς το πλέον σημαντικό πρόγραμμα ε, μεταρρύθμισης του διεθνούς επενδυτικού ε, συστήματος. Ας δούμε τώρα τι έχουμε κάνει εσωτερικά. Όπως θα γνωρίζετε, στη δέσμη ε, εμπορικών μέτρων ε, της ε, κατάστασης της Ένωσης ακούσαμε για μια σύσταση να εξουσιοδοτηθεί η Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις έχουμε υιοθετήσει στο πλαίσιο αυτό σχέδια διαπραγματευτικών εντολών. Όπως θα γνωρίζετε, οι οδηγίες αυτές μαζί με τις οδηγίες ε, για τις συμφωνίες με την Αυστράλια και την Νέα Ζηλανδία είναι οι πρώτες που δημοσιοποιούνται αμέσως μετά από την υιοθέτησή τους από τους επιτρόπους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και με οδηγεί στις επόμενες παρατηρήσεις μου στο ότι στα επόμενα μου σχόλια το πόσο ε, σημαντική βλέπει η Κομισιόν τη διαφάνεια σε τέτοιου είδου προγράμματα. Τα έγγραφα αυτά λοιπόν εγκρίθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με αυτά προτείνεται οι διαπραγματεύσει να λάβουν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη. Θα σας το περιγράψω πιο λεπτομερώς αργότερα προτείνουν επίσης μια ε, διεπίπεδη δομή ε, δικαστηρίου με δικαστές πλήρους απασχόλησης όπως είπα. Επίσης αναφέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη θέση των αναπτυσσόμενων χωρών και των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών εντός του συστήματος. μια ιδέα όλο και πιο δημοφιλή όσον αφορά τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι να δημιουργηθεί ένα κέντρο συμβουλευτική υποστήριξη το οποίο θα προσφέρει αρρωγή στι αναπτυσσόμενε και λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε ε, όταν πρέπει να ασχοληθούν με ε, υποθέσει ε, διαφορών στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση της σύστασης και των οδηγιών, δημοσίευσαμε και την εκτίμηση δικτύπου που πραγματοποίησε η Κομισιόν το τελευταίο έτος. Αυτή είναι η πρώτη λεπτομερή εκτίμηση δικτύπου που αναλύει το ενδεχόμενο δημιουργία ενό επενδυτικού δικαστηρίου. Περιλαμβάνει ανάλυση των πιθανών κόστου ενό πολυμερού επενδυτικού δικαστηρίου, γιατί είναι και πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Και αυτά τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου, Φυσικά ήρθαμε σε τακτική επαφή με ενδιαφερομένους. Είχαμε μια συνάντηση με ενδιαφερομένους που έγινε το Φεβρουάριο με την κυρία Μάλμστρομ το... σχετική μαγνητοσκόπηση υπάρχει διαθέσιμη online. Πραγματοποιήσαμε μια δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου. Εκεί λάβαμε πολλές απαντήσεις οι οποίες αναλύθηκαν και έχουν ληφθεί υπόψη στην εκτίμηση αντικτύπου. Η επαφή μας με τους ενδιαφερομένους συνεχίζεται. πρόκειται να οργανώσουμε μια συγκεκριμένη ε, συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών για τα ζητήματα αυτά στις 20 Νοεμβρίου και θα συνεχίσουμε να έχουμε τακτικές συναντήσεις με διαφόρους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή. Και φυσικά υπάρχει και μια ειδική ε, ιστοσελίδα με πληροφορίες για το έργο αυτό. Τώρα θέλω να σας ε, κάνω μια σύντομη περιγραφή των εξωτερικών εξελίξεων. τον Ιούλιο φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κρατημέλη της, ο Καναδάς και κάποιες άλλες χώρες ε, ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να ξεκινήσουν τις εργασίες επί του θέματος αυτού. Από τον Νοέμβριο και μετά η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών, η UNCITRAL, θα ξεκινήσει τις εργασίες της για να συζητήσει τη συνολική μεταρρύθμιση του ε, καθεστώτος ε, επίλυσης διαφορών σε εμπορικά θέματα και σε επενδυτικά θέματα, συγγνώμη. Γιατί θεωρούμε ότι η Uncitral είναι το καλύτερο φόρουμ για τις συζητήσεις αυτές. Ε, ένα αδιάστο επιχείρημα είναι ότι είμαστε πεπισμένοι ότι για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο, πρέπει να είναι πραγματικά πολυμερές. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι απολύτως ανοιχτή σε όλους τους φορείς και το πλεονέκτημα της διαδικασίας ε, στο πλαίσιο της Ονσιτρέλ είναι ότι όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών ε, και οι παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών καθώς και οποιαδήποτε ενδιαφερόμενα μέρη είναι δυνατόν να συμμετάσχουν. Δηλαδή και οι διεθνείς οργανισμοί ε, ε, τους οποίους αφορά το ζήτημα Η κοινωνία των πολιτών επίσης ε, μπορεί να διαπιστευτεί και να συμμετέχει στις συζητήσεις. Ε, θεωρούμε επίση ότι η Ονσιτράλ είναι το καταλληλότερο φόρουμ λόγω της εκτενούς διαφάνειας που παρέχει. Η, τα πρακτικά των συναντήσεων δημοσιοποιούνται άμεσα, οι ε, ηχητικές μαγνητοσκοπήσεις είναι διαθέσιμες άμεσα, οπότε όποιος από εσάς έχει χρόνο αργότερα μπορεί να ακούσει ε, πενθήμερες συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του ΑΕΣΔΙΕΣ από ηχητικά αρχεία. Τον Ιούλιο φέτος τα Ηνωμένα Έθνη ε, έδωσαν τρεις συγκεκριμένες εντολές ε, στην αρμόδια ομάδα εργασίας. Η μία εντολή είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη να διασφαλιστεί ότι οι συζητήσεις θα γίνουν μεταξύ όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων ε, συγκεντρώνοντας πολλού και διάφορου ενδιαφερομένου και ειδικότερα από ε, κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις. Το άλλο στοιχείο της εντολή είναι το εξής. Κάτι που εμείς έχουμε αναγνωρίσει είναι ότι δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσμου τις συζητήσεις που είχαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για τις επενδυτικές πολιτικές τα τελευταία χρόνια. Πολλές έχουν κάνει συζητήσεις, αλλά ε, οι οποίες δεν προχώρησαν τόσο όσο προχώρησαν οι συζητήσεις μας. Κατά συνέπεια κατέστησα φέσο ότι η ομάδα εργασίας ε, θα πρέπει να ε, διέλθει από τρία βήματα για να μπορέσει να προχωρήσει τις εργασίες της. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσδιορίσει και να εξετάσει τις ανησυχίες όσον αφορά το ISDS. Μετά θα πρέπει να αναλύσει το είδους μεταρρυθμίσεις είναι επιθυμητές. Και τρίτον, θα χρειαστεί να ε, εκπονήσει λύσεις ε, για να... τα προβλήματα αυτά. Αυτά είναι τα τρία σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η ομάδα εργασιών. Η πρώτη συνέντευξη της ομάδας εργασιών θα λάβει χώρα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου στη Βιέννη. Προ ενημέρωσή σα υπάρχουν εδώ συνδέσει προ τα διάφορα έγγραφα τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα για τη συνεδρίαση αυτή. Μια δεύτερη συνάντηση θα λάβει χώρα 23 έως 27 Απριλίου του 2018. Αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη για να συνεχίσει τις εργασίες ε, επί της εντολής αυτής και τον Ιούλιο του χρόνου η ομάδα εργασίας θα εκπονήσει έκθεση προς την, ε, UNCITRAL, ε, προς την Επιτροπή UNCITRAL και ναι, να αναμένεται ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά πρόκειται για ένα φόρουμ το οποίο θα συζητήσει την ε, συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης επενδυτικών διαφορών και την ενδεχόμενη σύσταση ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου. Κομισιόν είναι ιδιαίτερα δραστήρια ε, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων ε, που έχουν εκφράσει ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Μάλμστρομ για την πρωτοβουλία αυτή. Οπότε πολλαπλησιάζουμε τις επαφές μας. Ε, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η κυρία Μάλμστρομ μίλησε σε ένα σεμινάριο στη Σεούλ το Σεπτέμβριο όπου συμμετείχαν πολλές ε, χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή ε, μαζί με διάφορους ακαδημαϊκούς ε, και ακολούθησε κάποια συζήτηση των θεμάτων αυτών με πολλές χώρες από την περιοχή της Ασίας. Στις αρχές της εβδομάδας αυτής ήμασταν στα Ηνωμένα Έθνη σε μια διασκέψη για το εμπόριο και την ανάπτυξη στην ετήσια διάσκεψή τους Συζητήθηκε η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Επενδυτικού Συστήματο και η ιδέα του πολυμερού δικαστηρίου είναι κάτι που έχουμε προτείνει εμεί και το οποίο δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης ε, θα συνεχιστούν διάφορε ad hoc άτυπες συζητήσεις ε, στο όρατο μέλλον σε... ταυτόχρονα με τις εργασίες της ε, UN Central. Κύριε Πρόεδρε, εδώ ολοκληρώνονται οι παρατηρήσεις μου. Φυσικά η Κομισιόν με μεγάλη ευχαριστήση θα απαντήσει σε οποιασδήποτε ερωτήσει έχετε, η σχόλια. Επίσης με μεγάλη μας χαρά θα σας κρατήσουμε ενήμερος καθώς θα προχωρούν οι συζητήσεις ε, στην ε, UNCTRAL μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δέκα συνάδελφοι θέλουν το λόγο και έχουμε 20 λεπτά. 1,5 λεπτό ο καθένας λοιπόν. 90 δευτερόλεπτα. Η κυρία Κέρτον Darling. Ευχαριστώ. Πολλά χρόνια συζητάμε αυτό το θέμα Colin και χαιρετίζω αυτή την αλλαγή στάσης της Κομισιόν δεν είχαμε πάντα την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοούσε την ανάγκη αλλαγής της επενδυτικής μας πολιτικής. Σημειώνω λοιπόν αυτή την ε, ευπρόσδεκτη αλλαγή. Ερωτήσεις. Λόγω αυτής της αλλαγής θα υπάρξει ένα μορατόριο στην διαπραγμάτευση διμερών επενδυτικών συμφωνιών μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση για το πολυμερές δικαστήριο και για τις αρχές που θα το διέπουν. Κατόπιν, μια σειρά από χώρες στον κόσμο μονομερός εγκαταλείπουν διμερείς εμεδυτικές συμφωνίες σε η Νότια Αφρική, η Ινδία και άλλες. Ποια είναι η στάση της Επιτροπής προς αυτές τις χώρες, ε, τι κίνητρα θα τους δώσουμε για να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια για ένα πολυμερές δικαστήριο. Τρίτον, τα καθήκοντα των επενδυτών. Πάντα ήμασταν σαφείς. Έχουν δικαιώματα οι επενδυτές, αλλά έχουν και υποχρεώσεις, καθήκοντα, καθήκοντα έναντι των χωρών στις οποίες επενδύουν. Πώς θα λειτουργήσει. Θα πρέπει να έχει σεβαστεί κανεί, για παράδειγμα, ε, τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικαστήριο. Μόνο οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση στο δικαστήριο ή και ορισμένοι που έχουν ε, αιτήματα έναντι των επενδυτών. Ο κύριος Κέλλη Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αλλά χαμογέλασα όταν άκουσα στο 11.3 την ε, γραφειοκρατική διατύπωση. Αν η ομάδα εργασία θεωρήσει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση κλπ. κτλ. Μα δεν πρόκειται να καταλήξουν ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Αλλιώς ε, τι ρόλο θα παίζαν. Οπότε, οι λύσει τι οποίε θα καταλήξουμε και η δημιουργία αυτού του πολυμερού δικαστηρίου θα καταργήσουν τις αντιρρήσει ε, που τόσο έντονα εξέφρασαν πολλοί ότι δεν μπορούν να ε, στηρίξουν την ΣΥΤΑ, το TTIP, το Α, το άλλο κτλ. λόγω του παλιού μηχανισμού επίλυσης ε, διαφορών ούτω ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε εμπορικέ συμφωνίε χωρί να έχουμε αυτό το αγκάθι. Ευχαριστώ πολύ η Καρολίν. Ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετίζω αυτή τη μεταρρύθμιση. Είναι σημαντικό ότι θα έχουμε τώρα δημόσιο, όχι ιδιωτικό δικαστήριο. Ερωτήσεις. Αυτό το νέο πολιετές επενδυτικό δικαστήριο, ποιος θα μπορεί να απευθύνεται σε αυτό. Θα έχει ειδικό δικαίωμα μια πολυεθνική. Αν θέλουμε ίση μεταχείριση, τι θα γίνει με τους πολίτες ή με τους επενδυτές, ε, τους εγχώριους από μια χώρα. Και τι θα γίνει με το ρόλο της εθνικής δικαιοδοσίας. Δεν θα πρέπει πρώτα αυτοί να εξαντληθούν, να εξαντληθούν δηλαδή οι προσφυγέ αυτού και μετά να μπορεί να προσφύγει κανείς στο πολυμερές αυτό δικαστήριο. Και τρίτη ερώτηση. Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας για τους δικαστές αυτού του δικαστήριου, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν αναγκαίος. Σούστα. Ναι, παρόμοιε ερωτήσει κατά τη συζήτηση για αυτό το δικαστήριο και την προστασία των επενδύσεων. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν ότι δίδουμε μόνο δικαιώματα στους επενδυτές και δεν τους επιβάλλουμε υποχρεώσεις. Ποια θα είναι η νομική βάση του δικαστηρίου αυτή, τι υποθέσεις θα μπορεί να εξετάσει. Για παράδειγμα, τα κεφάλαια βιωσιμότητας δεν θα μπορούν να ε, είναι αντικείμενο προσφυγών εάν κάποιοι επενδυτές δεν τα τηρούν. Η Τιτσιάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι και πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την πρόταση. Φαίνεται σύγχρονη και διαφανής ε, η πρόταση της Κομισιόν, ωστόσο πιστεύω ότι είναι μια ε, απελπισμένη προσπάθεια να επενεργοποιήσει το ISDS που θα βοηθά ομίλους να κάνουν μηνύσεις σε κράτη. Οπότε παραμένουν κάποια σημεία πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου που είναι ανεπίλητα χρειαζόμαστε. Ε, είναι ένα μονοκατευθυντικό σύστημα. Μόνο οι πολυεθνικοί μπορούν να κάνουν μηνύσεις σε κράτη, όχι το αντίστροφο. Και δεύτερον, δεν επιτρέπει να εξαντληθούν όλα τα δικαστικά επίπεδα πρώτα απ' όλα και δεν εξετάζει επίσης τη συγκρούση συμφερόντων των δικαστών. Επίσης, όπως και άλλα δικαστήρια υπάρχει κίνδυνος ε, να επεκταθούν και σε άλλους τομείς που δεν εντάσσονται στην επίλυση επενδυτικών διαφορών. Είναι φυσιολογικό ένα δικαστήριο να θέλει να διευρύνει ε, το πεδίο αρμοδιοτήτων του ε, και να καταπατήσει αρμοδιότητες κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκ των πραγμάτων διεθνείς επενδυτές και όμιλοι θα έχουν περισσότερα προνόμια από πολίτες και κράτη. Ειλικρινά λοιπόν θεωρώ ότι δεν μιλάμε εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις μεγάλες πετρελαϊκές ε, ε για να μειώσουμε το κόστος των ε, ε, φαρμάκων και των δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις μεγάλες υπηρεσίες και τους μεγάλους ομίλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος Μπούχναρ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις ερωτήσεις που υπέβαλαν ε, οι προηγούμενοι ομιλητές. Τα κράτη θα μπορούσαν να προσφύγουν κατά των πολυεθνικών. Δεν είναι μόνο για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και για κοινωνικά θέματα και για άλλες ρυθμίσεις και κανόνες των κρατών. Πρόκειται για φυσιολογικούς και κανονικούς κανόνες που εφαρμόζουν τα κράτη. Αν δεν τηρούνται θα πρέπει να μπορούν να προσφύγουν. Γιατί είναι πολύ περιορισμένη από ό,τι φαίνεται η δυνατότητα προσφυγή των κρατών. Είναι δυνατόν να διευρυνθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουταλα. Είναι ένα βήμα πρόοδου. Μια θεσμική πρόοδος για τη ρύθμιση διαφωνιών. Αλλά ακριβώς υπάρχει το θέμα που έθεσε η συνάδελφος Κέρτον Ντάρλιν. Υπάρχει θέμα εξισορρόπησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επενδυτών και κατόπιν. Πώς, για παράδειγμα, θα εφαρμόζεται η τήρηση των κεφαλαίων βιώσιμης ανάπτυξης. Να δούμε πώς θα τα πάει η αναθεώρηση της Συμφωνίας Ένωσης Καναδά. Και υπάρχει και το θέμα που έθεσε η κυρία Φορέντσα. Θα πρέπει να υπερτερούν οι διεθνείς συμφωνίες, όπως η Συμφωνία του Παρισίου, οποιασδήποτε αλλη ε, αποφαση Πώς λοιπόν θα μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να μας δώσει αξιόπιστες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Βιβιάννα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά του ΕΛΚ και με τη συμφωνία της συντονίστριάς μας, της κυρίας Βουιθφολτ, πρέπει να πω ότι μας ικανοποιεί ότι τη μέρα που θα γίνει ψηφοφορία για την ενδυνάμωση των μέσων εμπορική άμυνας υποβάλλονται και αυτές οι προτάσεις για ένα πολυμερές δικαστήριο. Ορίστε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που μας βρίσκουν συμφώνους. Και, όπως λέει η Γκοτλίβ, είχαμε συντάξει την τροπολογία του Μαρτίου 15 και τώρα, δυόμιση χρόνια αργότερα, βλέπουμε τι έχει γίνει. Τότε η συζήτηση ήταν για το TTIP και το ISDS. Τώρα έχουν αποσυρθεί και τα δύο. Άλλαξε λοιπόν η κατάσταση θετικά. Κινούμεθα προς μια ανοιχτή και διαφανή κατεύθυνση με μία ε, προβλέψιμη νομολογία. Ακριβώς αντίστροφη είναι η κατάσταση από την κατάσταση όπως ήταν τότε που υποβάλαμε την τροπολογία μας. Αλλά τα δύσκολα είναι ακόμη μπροστά μας. Θα μας στηρίξουν οι Καναδοί, οι Βιετναμέζοι και διάφοροι άλλοι. Το δικαστήριο αυτό θα έχει αρμοδιότητα για όλες τις διμερείς συμφωνίες επενδύσεων που έχουν ε, ε, υπογράψει τα κράτη-μέλη. Θα καλύπταμε τότε τις μισές εμπορικές συμφωνίες που υπάρχουν στον κόσμο, 1.400 από τις 3.000. Και τι γίνεται στο Συμβούλιο. Ποιος φρενάρει, ποιος θέλει να υπάρξει θετική λύση, τι εταίρους έχουμε στον κόσμο, ποια είναι η γνώμη τους τι συμμάχους θα έχουμε, με ποιους πρέπει ακόμη να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ιωάνν Μαρή Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα είμαι σύντομη. Καταρχάς, κάποιες ε, συμφωνίες ε, ε, στο παρελθόν Μπορεί να γίνονται ακόμη και σε δωμάτια ξενοδοχείου. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν ήταν αυτό με το ISTS. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν πολλές αντιρρήσεις για το ότι οι πολυεθνικές θα μπορούσαν να προσφύγουν κατά κρατών που θα είχαν λάβει ε, δημοκρατικές αποφάσεις, δηλαδή αποφάσεις με βάση την ε, δημοκρατική του ενωμή τάξη. Έχουμε τι περιπτώσει τη Γερμανίας, ε, του Εκουαδόρ, της Ρουμανίας. Μπορεί και με το νέο σύστημα να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτή η ιστορία να μην γίνονται σε γωνίες και σε δωμάτια ξενοδοχείων αυτές οι διαδικασίες, ε, εντάξει είναι θετικό, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι προσβολή προς την νοημοσύνη όσων ε, κατά την δημόσια διαβούλευση εκφράστηκαν κατά του ISDS. Τι προστιθεμένη αξία θα μας δώσει αυτό το δικαστήριο. Τι περισσότερο έχει να μας προσφέρει έναντι για παράδειγμα των ε, διαιτητικών μηχανισμών του ΠΟΕ ή των δικαστηρίων. Και γιατί διαλέξαμε την Ούμου Σιτράλ και όχι κάποιο άλλο φόρουμ για να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να εξαντληθούν οι εθνικές δυνατότητες ε, δικαστικής επίλυσης πριν στραφούμε σε αυτό το δικαστήριο. Θα έπρεπε λοιπόν πάντα να εφαρμόζεται πρώτα η εθνική νομοθεσία για αυτές τις συμφωνίες. Τι θα κάνετε για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, για παράδειγμα, υπάρχουν ε, δυνατότητες προσφυγής ε, σε, ε, στις ασφαλιστικές εταιρείες και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών, SSDS. Αυτό το νέο σύστημα δίνει δυνατότητα να προσφεύγει ε, μία πολυεθνική κατά κρατών. Αλλά ποιοι άλλοι θα μπορούν να προσφύγουν. Όλα αυτά είναι αδικίες. Και τι ρόλο θα παίξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα υπάρξει κάποιο ψήφισμα. Ο Χέλμουντ Σόλτς. Θα είμαι σύντομο. Γιατί πολλά υπόθηκαν. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει τι προτεραιότητα και τι κατάταξη θα υπάρχει. Και σε τι πλαίσιο θα λειτουργήσει. Δεν είναι στα πλαίσια του ΟΗΕ, θα αναπτυχθεί περισσότερο εντός του ΠΟΕ. Πώς βλέπει τις σχέσεις που θα έχει ο ΟΗΕ και ο ΠΟΕ με αυτό το δικαστήριο η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος εγώ, Κόλλιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει μόνο μία συμφωνία που να περιέχει το παλιό σύστημα ISDS. Είναι η ενεργειακή χάρτα. Δεν είναι λογικό τώρα η Επιτροπή να προτείνει ένα νέο σύστημα που θα αλλάξει και την ενεργειακή χάρτα για να την εντάξει στο νέο σύστημα. Παρακαλώ, Κόλλιν, πες μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για το ενδιαφέρον και για τα σχόλιά σας. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αλλά και πιο απλά. Καταρχάς δύο βασικές παρατηρήσεις. Στόχος μας εδώ είναι να αντικαταστήσουμε το υφιστάμενο ISDS, Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτή και Κράτους. Στόχος δεν είναι να αλλάξουμε τους υφιστάμενους κανόνες. Η δουλειά για τη μεταρρύθμιση των κανόνων γίνεται μέσα σε άλλους μηχανισμούς, τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών ή άλλους μηχανισμούς γενικότερα, αλλά στόχος μας δεν είναι να μεταρρυθμίσουμε τους κανόνες. Μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους διαδικαστικούς κανόνες και το είδαμε αυτό και στο ΠΟΕ. Όταν πρόκειται για την ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και εμπορίου ή εργασιακών προτύπων και εμπορίου, είναι καλό να έχουμε ένα μόνιμο σώμα που δίνει καλύτερα αποτελέσματα και υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πτυχών. Και άρα στόχος μας είναι και εδώ να πάμε προς μια παρόμοια παρεμφερή κατάσταση. Δεν είναι πρόθεσή μας να υπάρξει μορατόριου ε, των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών και των συμβάσεων. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί στις διμερείς συνθήκες προβάλαμε ένα ε, σύστημα διμερές δικαστικό επίλυσης διαφορών και όταν τα κράτη-μέλη ζήτησαν την έγκριση να διαπραγματευτούν, απαιτήσαμε να υπάρχει παραπομπή στο πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Άρα το ISDS θα αντικατασταθεί από το πολυμερές δικαστήριο και τη διαδικασία του όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα. Η κυρία Ρέντιμ και ο κύριος Κάρτον Ντάρλινγκ έθεσαν τα ίδια ερωτήματα πάνω κάτω και απαντώ λέγοντας ότι πολλές τρίτες χώρες ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως. Ο βαθμός ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν είναι διαφορετικός. Κάποιες χώρες ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως, κάποιες είναι απλά περίεργες και θέλουν να τα παρακολουθήσουν λίγο περισσότερο τα ζητήματα αυτά. Όλες οι χώρες συμφώνησαν στην εντολή που δόθηκε από τον κύριο Τσαόπ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας και τελικά και τον ΙΠΑ και, της, και την Ιαπωνία μετά από κάποιες περιπλοκές συζητήσεις. Όλες οι χώρες λοιπόν που παρέστησαν συμφώνησαν να δουλέψουν περαιτέρω στην παγκόσμια αυτή δουλειά μεταρρύθμισης για το ISTS. Δεν απαιτείται να αλλάξουν την πολιτική τους. Και το ISTS με το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο μεταρρυθμίστε λιγότερο από αυτά που προτείνουμε εμείς εδώ. Τα παρακολουθούμε λοιπόν όλα αυτά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Μεγάλο στόχο είναι να καλύψουμε τουλάχιστον τις 1400 συνθήκες και θέλουμε και η συνθήκη για την ενεργειακή χάρτα να καλυφθεί. Γίνονται επίσης συζητήσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένη συνθήκης για την ενεργειακή χάρτα και τη μεταρρύθμιση. Άλλα Άρα όλα βαίνουν προς την μεταρρύθμιση της συνθήκης για την ενεργειακή χάρτα. Τώρα για τη σχέση με τα εθνικά δικαστήρια. Αυτά, αυτός είναι ένας μηχανισμός διεθνούς επίλυσης διαφορών. Μπορεί να συγκριθεί με το ΠΟΕ, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με διάφορα άλλα φόρουμ όπου έχουμε διεθνείς κανόνες που τίθενται σε ισχύ από διεθνείς μηχανισμούς. Πολλά χώρια δικαιακά συστήματα δεν ενσωματώνουν αυτούς τους διεθνείς κανόνες στην εσωτερική ένωμη τάξη, άρα αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν είναι τουλάχιστον αδύνατο για τις διεθνές, διεθνείς συμφωνίες να αντιμετωπιστούν στα εθνικά δικαστήρια. Τα εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν αυτό το διεθνή μηχανισμό επίλυσης διαφορών και είναι σημαντικό η σχέση μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και διεθνών δικαστηρίων να γίνεται σεβαστή και μάλιστα σε διάφορες συνθήκες. Οι περισσότερες συνθήκες το αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Και αυτό πρέπει να συζητηθεί έτσι περαιτέρω καθώς θα προχωρούμε στις διαπραγματεύσεις για το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Πολλοί από εσά θέσατε το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τις υποχρεώσεις των πολυεθνικών και των επιχειρήσεων και των μεγάλων επενδυτών. Θα γνωρίζετε ότι στις συζητήσεις ε, λαμβάνουν χώρα διάφορες δράσεις και εξετάζονται διάφορα στοιχεία και ζητήματα Υπάρχει η δουλειά της ε, Επιτροπής για την εταιρική ευθύνη και υπάρχει αυτό στις συνθήκες. Πρόθεση της Επιτροπής, η δουλειά για την εταιρική ευθύνη και τις υποχρεώσεις του επενδυτή να συνεχιστούν, να αποτελέσουν σε σημαντικό βαθμό μέρος της πολιτικής και στο βαθμό που οι συμφωνίες αρχίζουν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των επενδυτών και υπό τον όρο ότι προβλέπονται αυτά από τις συνθήκες, τότε ναι και το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο θα μπορέσει να ε, δικάσει πρόσφυγες σε βάρος των επενδυτών. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν ε, αντεγκλήσεις και ε, counterclaim δηλαδή από πλευράς κρατών. Και δύο τελευταία σχόλια. Είμαστε στα αρχικά στάδια της συζήτησης στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές στηρίζει αυτό το project, αυτό είναι δίκαιο να το πει κανείς. Περιμένουμε σχετικά γρήγορα να προχωρήσει για να έχουμε συμφωνία για έγκριση τους επόμενους μήνες. Για το ερώτημα του κυρίου Σόλτς, πού όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν. Εμείς θεωρούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι το καλύτερο μέρος για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Εκεί μπορούμε να τους περιλάβουμε όλους, να έχουμε όσο το περισσότερη διαφάνεια και ούτω καθεξής. Άλλο τώρα είναι πού τελικά θα έχει έδρα το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Στο ΠΟΕ είναι μια επιλογή. Αλλά μάλλον είναι απίθανο έτσι όπως έχει ο ΠΟΕ αυτή τη στιγμή, σε βραχυπρόθεσμη βάση τουλάχιστον. Μια επιλογή είναι ο ΠΟΕ, ίσως άλλα μέρη, άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Μπορεί τελικά αυτός ο θεσμός να γίνει ένας θεσμός standard law, όλα αυτά θα τεθούν του. Ελπίζω να έχω απαντήσει. Ευχαριστώ, ο πρόεδρος. Και όσας ευχαριστώ, είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνουμε σε επαφή. Είναι κάτι που θα υποβάλει δηλαδή κανείς την προσφυγή του. Ελπίζω να έχω απαντήσει. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος και όσο σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνουμε σε επαφή. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Συγγνώμη Πρόεδρε να διακόψω ε, το φίλο που πήραμε μας λέει ότι μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν είναι καθόλου ευανάγνωστη η αναγραφή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και η διεύθυνση της ιστοσελίδας. Δεν μου απάντησαν στις ερωτήσεις μου και γι' αυτό θέλω να ψάξω στο διαδίκτυο τις απαντήσεις και δεν έχει καλά ε, τυπωθεί η διεύθυνση. Ναι, θα σας το δώσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα παραμείνουμε σε επαφή Είμαι πεπισμένος ότι και το Κοινοβούλιο θα κάνει δήλωση για το θέμα αυτό και πρέπει να δούμε με ποια μορφή θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πριν να υιοθετηθεί η εντολή από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Και δίνω αυτή αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Σαβή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης αυτό αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εργάζεται συχνά μελετώντας τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές δεδομένων των ζημιών που προκαλούν στους καταναλωτές και ε, των απολειών θέσεων εργασίας που δημιουργεί αυτή η πρακτική ως ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να έχουμε αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εμπορική πολιτική ασχολείται με το ζήτημα αυτό, το οποίο αποτελεί και προτεραιότητα της εμπορικής στρατηγικής του 2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο πρόσφατα. Η Επιτροπή σε έγγραφα που σχετίζονται με τη διθάσευση της παγκοσμιοποίησης ασχολείται επίση με αυτό το ζήτημα. Η εμπορική πολιτική πρέπει να προβλέπει κανόνες δίκαιους και ισότιμους για όλους τους φορείς. Έτσι θα πρέπει να αναπτυχθούν ορισμένα εργαλεία και κάποιες αρχές Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το σχέδιο γνωμοδότησής μου, όπου κάνω έκκληση για εξυγχρονισμό των εργαλείων εμπορικής άμυνας χωρίς να αποδυναμώνονται. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσουμε το κομμάτι της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του dumping, ώστε να επικαιροποιηθεί, γιατί τη στιγμή που υποβλήθηκε αυτό το κείμενο δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία για το θέμα αυτό. Ε, στο πλαίσιο τη καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού, επιμένω να υπάρχει αμοιβαιότητα να γίνει κεντρικό κομμάτι της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης ώστε να έχουμε και μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις αγορές των εταιρών μας. Είναι σημαντικό επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προωθήσει παγκοσμίω και στον ΠΟΕ τους κανόνες ε, θεμητού ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ευαισθησίες συγκεκριμένων τομέων. Τέλος, το σχέδιο γνωμοδότησης περιλαμβάνει πολλά σημεία που αφορούν συγκεκριμένα την αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν ζητήματα ανταγωνισμού στις εμπορικέ συμφωνίες και να διασφαλίζεται η τήρησή τους, στην προσοχή που πρέπει να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το θέμα αυτό και στο πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική και εναρμονισμένη τελωνιακή έλεγχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι τώρα ε, για τους σοσιαλιστές ε, Τζουτ Κεντάιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαφάη, την ε, εισηγήτρια, γιατί τη δημιούργησε μια πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Ε, επισημαίνει πολύ σωστά ότι χρειαζόμαστε ανταγωνισμό, ανταγωνιστική πολιτική για να καταπολεμήσουμε το αθέμητο εμπόριο. Κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση. Το δίκαιο εμπόριο μπορεί να προκύψει μόνο από δίκαιο ανταγωνισμό και οι κανόνες και οι κυρώσεις πρέπει να είναι ίδιες για όλους. Η Επιτροπή το αναγνωρίζει αυτό. Έχει κάνει κάποιε προσπάθειες ενίσχυση τη συνεργασία με τι ανταγωνιστικές αρχέ παγκοσμίω. Επίση, έχει συμπεριλάβει κάποιε διατάξει για τον ανταγωνισμό σε τελευταίε FTA. Αυτέ οι προσπάθειε κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να το αναγνωρίσει και η Κομισιόν. Η διεθνή συνεργασία δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε δομημένου μηχανισμού διασφάλιση τη ανταλλαγή πληροφοριών ή ευθυγράμμιση των πρακτικών. Κάτι το οποίο εμεί θα πρέπει να ενθαρρύνουμε για τι FTA. Έχουμε περιορισμένε διατάξει μέχρι στιγμή ε, με ελάχιστα μέσα εφαρμογή του. Κάτι που θα ήταν χρήσιμο, ωστόσο, πιστεύουμε, να ε, περιγραφεί καλύτερα στη γνωμοδότηση. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες για αυτά τα ζητήματα και αναμένω τη συνεργασία με τους σκιώδες. Ευχαριστώ. Για το ECR, ο κύριος Λούνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια και για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ε, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές. Καλό που είναι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει επιτέλους προσοχή στην ανταγωνιστική πολιτική ώστε να προωθήσουμε μια κουλτούρα ίσων συνθήκων ανταγωνισμού. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Θέλω να θέσω ορισμένα συγκεκριμένα σημεία τώρα. Αυτό που θέλουμε εμείς να περιλαμβάνει αυτή η έκθεση είναι να ενδυναμωθεί η πολιτική ανταγωνισμού ε, ως προς την Ασία Πολύ συμφωνούν μαζί μου νομίζω γι' αυτό και να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ αρχών ανταγωνισμού. Το ιδανικό θα ήταν η συνεργασία αυτή να είναι παγκόσμια, ώστε να υπάρχει συνοχή παγκοσμίω. Επίσης ε, θα ήθελα να δω μείωση ε, του κόστους της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Όπως ξέρετε έχουμε αυτές τις, ε, τη συμφωνία δεύτερης γενεάς ε, μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που συνάφθηκε το 2013. Πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά για να δούμε πώς μπορούμε να αποκομίσουμε κάποιες ιδέες. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις κρατικές επενδύσεις. Συμφωνούμε με την αρχή, ναι πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά αυτές ε, δεν πρέπει να μετατραπούν σε προστατευτισμό. Ειδικότερα δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να προσελκύσει ε, ξένες επενδύσεις ε, στα κράτη-μέλη. Για να γίνει κάτι τέτοιο δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι η γνωμοδότηση είναι πολύ καλή βάση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Θα κάνω δύο σχόλια. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ταχύτατες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Ε, οι ψηφιακές διαδικασίες κατακρεματίζονται ε, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και έχουμε και τις ε, διάστητες εκτυπώσεις τώρα. Ε, για παραδείγμα που ανατίθενται ξέρω εγώ, στην Ινδία και το προϊόν τελικά αποστέλλεται στις κατοχώρες. Όλα αυτά επηρεάζουν το διεθνή ανταγωνισμό. Ήθελα να πω λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιε είναι οι συνέπειε τέτοιων ε, εξελίξεων ε, στην απασχόληση στι χώρε μα, ειδικότερα στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, ατομικών επιχειρήσεων επίση. Οι οποίε απαιτείται να ανταγωνιστούν, καλούνται να ανταγωνιστούν με επιχειρήσεις άλλων χωρών. Ευχαριστώ πολύ για το ΙΕΝΕΦ, η κυρία Ζαμέ. Θα σας πω την απόψή μου για τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ΙΝΤΑ. Βλέπω υπάρχει μια τεράστια λίστα καλών προθέσεων, όπως αναφέρατε προηγουμένως καλό θα ήταν. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακριβώς το αντίθετο. FTA ανοίγεται σε αθέμητο ανταγωνισμό, σε ε, κακή ποιότητα προϊόντα. Ξέρετε, ούτε ο ανταγωνισμό, ούτε η εργασία και η νομοθεσία, ούτε οι κανόνε ασφάλεια ε, και περιβάλλοντο ε, δεν λειτουργεί τίποτα. Δείτε του ε, αποσπασμένου εργαζομένου. Τίποτα δεν λειτουργεί. Όταν μα λέτε να τηθασεύσουμε την παγκοσμιοποίηση, λαμβάνοντα μέτρα για να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών που απλά εντείνουν την παγκοσμιοποίηση. Τώρα, όσον αφορά τον ίσο ανταγωνισμό, εσεί ουσιαστικά εσκεμένα κάνετε ότι δεν βλέπετε το dumping που ασκείται εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της ε, μέσω του εμπορίου με ορισμένε τρίτες χώρες που υπονομεύει τον ανταγωνισμό. Επίσης ε, κλείνετε τα μάτια ε, στις φρικτές συνθήκες παραγωγής ορισμένων προϊόντων στην Ινδία, στον Παγκλαντές, στην Κίνα κτλ. Ο εξυγχρονισμός λοιπόν των μέσων εμπορικής άμυνας ε, θα έπρεπε να μας, ε, θα μας οδηγήσει σε μια ε, πολιτική πιο φιλελεύθερη. Τώρα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, πού είναι η αμοιβαιότητα στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΣΕΤΑ για παράδειγμα ζητήσαν τους Καναδούς να υιοθετήσουν καλύτερα πρότυπα περιβαλλοντικά ή υγειονομικά στα οποία υποβάλλουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Επίσης δεν μας λέτε τίποτα για την αμοιβαιότητα των αγορών ε, κινέζικων προϊόντων όπου η χνηλασιμότητα είναι 0 Περνώ στο σημείο 6. Μας λέτε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε όλοι εδώ ότι αυτοί που κερδίζουν από τις ε, ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών είναι οι πολυεθνικές, εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χωρίς καμία πραγματική πολιτική θεμητού ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε και για τη βούληση που υπάρχει όσον αφορά ε, τους αποτελεσματικούς και εναρμονισμένους ε, ε, τελωνιακούς ελέγχους του σημείου 7 να υπενθυμίσω ότι αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός νομιμοποιείται απόλυτα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών. Στο 8 μιλάτε για κανόνες αθέμητου ανταγωνισμού και θεμητού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Μιλάτε για ευαισθησία συγκεκριμένων τομέων, στους οποίους αναφέρθηκε χθε η Γεωργία. Μα έχετε αφήσει άναυδους. Ουδέποτε ε, προστατεύτηκαν οι γεωργοί μας μέχρι σήμερα η ΠΑΚΑ, ε, η ΣΕΤΑ και οι επακόλουθε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών κατέστρεψαν ε, πολύ ευαίσθητους τομεί όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλία. Επαναλαμβάνομαι γιατί, διότι πίσω από όλα αυτά, ξέρετε, υπάρχουν άντρες, γυναίκες που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς με τη δουλειά τους. Απλά ακολουθείτε μια πολιτική διανομέων εις βάρος των παραγωγών. Ε, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της και για την έκθεση που καλύπτει όλες τις πλευρές ε, του θέματος. Ήθελα απλώς να τονίσω ότι κάποια σημεία θα πρέπει να τονιστούν περισσότερο όπως το θέμα της αμοιβαιότητας γιατί κάτι που περιορίζει τον ανταγωνισμό είναι η έλλειψη αμοιβαιότητας ο διαφορετικές ερμηνείες των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ε, αμοιβαιότητα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στον ε, ισότιμο ανταγωνισμό και γενικότερα στις επιχειρήσεις. Κάτι άλλο. Η πρόσβαση στην ενέργεια ή σε διαφορετικές πηγές ενέργειας. Η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πηγές ενέργειας είναι επίσης ένα, ένα στοιχείο δίκαιο ανταγωνισμού. Και κάτι άλλο. Οι δημόσιες προμήθειες. Μία από τις δυνατότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν για να υψωθούν τύχη προστατευτισμού και για να περιορίσει κανείς την ε, πρόσβαση όλων στην αγορά είναι ο περιορισμός της πρόσβασης ε, στους δημόσιους διαγωνισμούς. Και αυτό θα επιχειρήσω να το διορθώσω μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Σια Χένιγκ. Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε εδώ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, μαζί με τη συνάδελφό μου που θα απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσει. Ευχαριστώ τον για την εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση. Ορισμένα θέματα αφορούν τον ανταγωνισμό και ορισμένα αφορούν ε, το εμπόριο, αλλά φυσικά αυτά τα δύο δεν είναι ε, το ένα από το άλλο και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να τα εξετάζουμε ε, από κοινού και ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Ζαϊφή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ το σύνολο των συναδέλφων που πήραν τον λόγο. Σημείωσα τις παρεμβάσεις τους, τα επιχειρήματά τους. Εδώ και χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι το θέμα αυτό έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Θα πρέπει λοιπόν να αποτιμούμε σωστά την επίπτωση των αποφάσεων μας. Ε, το θέμα που θέσατε της αμοιβαιότητας για μένα ήταν ε, στο επίκεντρο των θεμάτων που ε, υπάρχουν και των επιπτώσεων κάποιων αποφάσεων. Σημειώνω λοιπόν αυτά που είπατε και θα αρχίσουμε τώρα την εργασία μας για αυτή την γνωμοδότηση ε, λίγα προσεχώς. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Προθεσμία για τροπολογίε. 17 Οκτωβρίου. 6 ώρα το απόγευμα. 17 Δεκάτου 18. 00. Οπότε, Κλείσαμε το σημείο 15 και δεν έχουμε καθυστέρηση. Σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει η περίοδος ψηφοφοριών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πριν αρχίσουμε το σημείο 16, σας παρακαλώ να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες σας. Βούντε λίμπε. Έρχεται η κάρτα μου. Εγώ όμως έχω φτάσει. Ναι, μα σε βλέπω. Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία. Hm. Δεν ψηφίσατε όλοι δεν βλέπουμε όλες οι κάρτες να χρησιμοποιήθηκαν. Για να δούμε. Όσοι έβαλαν τις ε, κάρτες τους στο μηχάνημα, όντως μετρήθηκε η ψήφος τους. Για να ξαναδούμε. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Πέρα τη δοκιμαστικής και σημειώνουμε ότι λείπει μία ψήφος. Λοιπόν, πρόταση διαπραγματευτικής εντολής για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την 22 άρχεται πέρας ψηφίσατε όλοι καλώς ωραία εγκρίνεται τροπολογία 26 26 υπέρ Όχι, 23 υπέρ παρακαλώ. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχουμε μια προφορική τροπολογία ως προσθήκη προφορική τροπολογία ως προσθήκη στην συμβαστική 5. βεβαίω, ακριβώ Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 86 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. 88 δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 88 άρχεται. πέρασε. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά δεν σας προλαβαίνουν ούτε οι διερμηνείους ούτε εγώ να γυρίσω τις σελίδες. Έλεος. Βεβαίω, πρέπει να τρώμε αργά και να ψηφίζουμε αργά. Μα δεν βλέπω φαΐ, λέει η κυρία Μακλάχλα. Ωραία. Οπότε, 107. 107 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά να επαληθεύσουμε. 108 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, να επαληθεύσουμε, ψηφίζουμε την 109. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 114. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 120. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβα... Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16α συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 16α συμβιβαστική. Πέρασε. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 159. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 167. Πέρασε. Απορρίπτεται.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 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Από την άγκρη τώρα. Άγκρι 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την τροπολογία της Άγκρι υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άγκρι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά. Ε, Άγκρι 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 της άγκρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 άγκρι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. κατά. Α, νέα συμμαχία βλέπω. Νέος συνασπισμός. Την ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 25 της Άγκρη. 25 από την Άγκρη. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Καλώς. Ψηφίζουμε το σύνολο τώρα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία. Πέρασε. Συγχαρητήρια με μεγάλη πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Αλλά δεν είναι εδώ ο εισηγητής. Αυτά με την Αυστραλία. Πάμε τώρα στο ίδιο εγχείρημα με την Νέα Ζηλανδία, αν δεν απατώμε. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30... 33 προέδρος, 30 πρώτα απ' Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές. Τι γίνεται με το EFTD για τη 46. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία για την συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72 είναι η επόμενη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά δεύτερο τμήμα της 91 να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 91 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 109 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 110 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 111 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ε, συμβεστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 129, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 149. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές άρχεται η ψηφοφορία για την 154 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε τροπολογία 8 άρχεται πέρας απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται, νομίζω. Σκόντε τα χέρια σας, α. Ε. Μην το ξεχνάτε. 16, υπέρ. 14 εγκρίθηκε. 16, υπέρ. Κατά. Τέλεια. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 20 άρχεται η ψηφοφορία And the vote is Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι ε, γνωμοδότηση άγκρι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την άγκρι 13 άρχιτη ψηφοφορία And vote is Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 16 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία Vote is closed. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. Άγκρι 17. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Συγγνώμη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Άγκρι 20. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Άγκρι 24. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την άγκρη 24 Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Άγκρη 26. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και για το ολοκείμενο ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και πάλι. Και πάμε στο σημείο 18. Ε, μιλάμε για το πνευματόδη του κυρίου Ντάντι. Πρώτη τροπολογία, υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Και η πράσινη. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη 37 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 και 40 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 41, 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το δούμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη 41. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 και 51 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι βέβαιος πολλοί δεν σήκωσαν το χέρι τους ε, ψηφίζουμε την 53η καλή προσπάθεια κύριε Τάκουλα πέρας εγκρίνεται έχετε δίκιο 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61-62 ταυτόσημες υπέρ κατά. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά να τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 61η και την 62η. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 σε 2 τμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα της 72ης τροπολογίας. Ξεκινάμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 και 85 ταυτόσημες τις ψηφίσουμε μαζί υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. 86 και 87 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. 88 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 και 94 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνονται.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 εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 και 33 και 34 βεβαίως του κυρίου Φίσας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και πάμε τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, με θαυμάσια μεγάλη πλειοψηφία, συγχαίρουμε τον κύριο Ντάντι για την υπερψήφιση της έκθεσής του. Ευχαριστούμε πολύ. So, we switch to number Τώρα περνάμε στο σημείο 19. Την τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα. Για τη νέα μεθοδολογία κατά του dumping. Έκθεση Τσίκου. Ευχαριστούμε τον συγκριτή. Νομίζω ότι έχουμε μια σειρά από νέα μέτρα που θα ασχίσουν παγκόσμια στην νομοθεσία κατά του dumping. Να ψηφίσουμε το κείμενο συνολικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται με ευρύτατη πλειοψηφία. Συγχαίρουμε τον συγητή. So, damit haben wir... Λοιπόν, τελείωσαν τις φορές. Σας ευχαριστώ πολύ για την θαυμάσια συνεργασία σας και να περάσουμε στο σημείο 20. Τώρα δεν είπα ότι πρέπει να αρχίσετε όλοι να φλιαρείτε. Απλώς είπα ότι περνάμε στο σημείο 20. Οι ομάδες ε, επιτήρησης. Έγιναν κάποιες συνεδριάσεις. Η πρώτη αφορά το Βιετνάμ. Έχουμε τον κύριο Ζαχραντήλ, τον θαυμάσιο συγητή μας και του δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από κάποια περίοδο διακοπής, ησυχία παρακαλώ. Excuse me. We relaunched the ξαναξεκίνησε η λειτουργία της ομάδας ε, επίβλεψης ε, για το Βιετνάμ γιατί πολύ σύντομα θα έρθει στην Επιτροπή μας η συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις με το Βιετνάμ. Είχαμε μια ευρία αντιπροσωπεία το Σεπτέμβριο πολυμελή από το εμπορικό ε, επιμελητήριο του Βιετνάμ συμμετείχαν και πολλοί άλλοι από τις χώρες ASEAN συμμετείχατε εσείς ως Πρόεδρος, ακούσαμε παρουσιάσεις από τον Γιέντ Ρίμπετ του Eurocham για την, το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο, ο οποίος μας έκανε μία παρουσίαση πολύ αναλυτική για την κατάσταση της οικονομίας του Βιετνάμ. Είχαμε επίσης τον επικεφαλή της διαπραγματευτικής ομάδας, τον κύριο Μάουρο Πετριτσόνε, έθεσε ορισμένα θέματα για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, ε, για το πώς θα καταλήξουν, καθώς και τον αντίκτυπο της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Και ακούσαμε μια παρουσίαση και του πρέσβη της Ένωσης στο Βιετνάμ, του κύριο Μπρούνο Άντζελεκ, που μας ενημέρωσε για την ε, τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Βιετνάμ. Για να δούμε τι στάση λοιπόν θα έχει και το Βιετνάμ για την εμπορική αυτή συμφωνία και την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω ότι τους προσεχείς μήνες ε, θα εντείνουμε την εργασία μας και θα καταφέρουμε κατά τη διάρκεια του επομένου έτους ε, να ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση για την ε, ε, εμπορική αυτή συμφωνία. Ο κύριος... Α, ο Πέδρο για την Ιαπωνία. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας συνεδρίασε στις 5 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουμε τη συμφωνία. Η κυρία Μάστρομ είχε έρθει εδώ στην Επιτροπή μας μετά τη συμφωνία επί της αρχής. Τώρα θα κάνουμε συζητήσεις ε, με τον Μάουρο Πετριτσόνε σε βάθος και με τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ένωση, τον κύριο Κοντάμα. Ξέρουμε ότι οι τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις θα συνεχιστούν και η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Παρά το ότι έχουμε εκλογές στην Ιαπωνία αλλά φαίνεται ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Τα κύρια θέματα που εξέτασε η ομάδα επιτήρησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ο μηχανισμός επίλυσης επενδυτικών διαφορών, διαφορών ε, επενδυτών και κρατών. Έχουμε μια σειρά από θέματα. Τονίσαμε την ανάγκη ε, να υπάρξει ένα εκτεταμένο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη για να μην απογοητευτούν οι προσδοκίες. Όπως ξέρετε, εμείς πιέζουμε πολύ για να δημοσιευθεί η εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές και χαίρομαι που τελικά το Συμβούλιο συμφώνησε να δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές το Σεπτέμβριο. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις 17 τρέχοντος μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ιγνάθιο, ευχαριστώ Πρόεδρε, για το Μερκοσούρ. Η ομάδα μας συνεδρίασε στις 7 ε, Σεπτεμβρίου. Εξετάσαμε το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, ε, μας τα εξήγησε η επικεφαλής ε, της διαπραγματευτικής ομάδας. Συναντηθήκαμε και Αργεντίνους βουλευτές από διάφορες ε, πολιτικές ομάδες. Μας εξήγησαν τις ανησυχίες τους, όπως και εμείς έχουμε τις δικές μας. Θέλουν να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση στη διαπραγμάτευση, να είναι πιο διαφανής. Και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση θα πρέπει αμφότερα τα κοινοβούλια να επικυρώσουν και να εξηγήσουν στους πολίτες το αποτέλεσμα. Χθες ε, σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ξέρουν ότι είναι σε κρίσιμη φάση διαπραγματεύσεις γιατί η Επιτροπή υπέβαλε την ε, προσφορά της για τα πιο επίμαχα θέματα Τονίζω λοιπόν ότι και το Κοινοβούλιο μας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις τελευταίες δύο εκφράσεις άποψης από αυτού του θέματος τόνισαν ότι πρέπει να είναι ισορροπημένη και αρμονική η συμφωνία που να εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Ένωσης και του Μερκοσούρ και ως Επιτροπή πρέπει να έχουμε επαρκή θεώρηση του θέματος αυτού για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα και να μην ε, περιοριστούμε σε κάποιους ε, κλάδους, όσο σημαντική και αν είναι. Έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, πρέπει να έχει ε, πρόσβαση στο εμπόριο αυτό και ο κόσμος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι θετικά τα πράγματα και θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές μας. Αυτό θα ωφελήσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της ομάδας επίβλεψης Mercosur για τη συμμετοχή του στην εργασία την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα. Θα έχουμε άλλη μια συνάντηση με την επικεφαλής της διαπραγματικής ομάδας για να δούμε πώς έχει πάει τελευταία, ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα στη Βραζιλία την προηγούμενη εβδομάδα και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 22 Νοεμβρίου σε ένα πιο γενικό επίπεδο. Ελπίζω να διευκρινιστεί καλύτερα η διάσταση της συμφωνίας αυτής. Ευχαριστώ πολύ όλους τους κοιόδης για τη συμμετοχή τους στις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Μαγρέμ. η κυρία Λαλόντ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οργανώσαμε μια συνεδρία παρακολούθηση 25 ε, Σεπτεμβρίου για το Μαγκρέμπ. Συζητήσαμε για το Μαγκρέμπ, για το Μαρόκο, για την Τινησία, για το Μαρόκο. Το θέμα ήταν να αξιολογήσουμε τις προόδους ε, του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κομισιόν και των Μαροκινών Αρχών που έλαβαν χώρα μέσα Ιουλίου. Όπως ξέρετε, πρόκειται να αλλάξουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης ε, Δεκεμβρίου του 2016 στην υπόθεση μεταξύ του Συμβουλίου με, με το μέτωπο Πολυσάριο. Εκτιμάται ότι είναι τρία ε, τα σημεία για τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε μια κοινή διατύπωση τροποποίησης της συμφωνίας. Ε, ένα κοινό κείμενο. Αυτό θα γίνει με μια ανταλλαγή επιστολών. Το δεύτερο θα είναι η αξιολόγηση των ωφελών της συμφωνίας για το λαό της Δυτικής Σαχάρας και το τρίτο είναι να έχουμε τη συνένεση του λαού από αυτά τα μέτρα. Η Κομισιόν μας είπε ότι έχει προχωρήσει στον πρώτο πυλώνα Ε, το CIA μα είπε ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο σημείο για το Μαρόκο, ότι η διαπραγμάτευση τη Συμφωνία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσει ε, την ειρηνευτική διαδικασία που αποτελεί το αντικείμενο διαπραγμάτευση. ταυτόχρονα στον ΟΗΕ. Θα υπάρξει συνεργασία με την Μάρτα Κόμπλερ, την ειδική δεταλμένη του ΟΗΕ. Μα είπαν ότι το εμπόριο με την περιοχή είναι περιορισμένο, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερε πληροφορίε για το θέμα. Μετά αναφερθήκαμε στην Τινησία με την οποία διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η Κομισιόν μας είπε ότι ο πρώτος γύρος ε, είχε καλή έκβαση. Αλλά ότι μετά η Τινησία επιβράδυνε την πρόοδο λόγω της νέας κυβέρνηση εν μέρη ε, στην Τινησία και λόγω των καθυστερήσεων ε, του πρώτου διαπραγματευτή. γίνεται μελέτη εκ των υστέρων ε, για την συμφωνία που υπήρχε. Θα παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις αυτές πολύ στενά και θα σας ε, κρατήσουμε ενήμερους για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τέλος Σιγκαπούρη, David Martin. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Η ομάδα παρακολούθησης ε, για τη Σιγκαπούρη έλαβε χώρα 26 Σεπτεμβρίου αξιοποιήσαμε την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού στις Βρυξέλλες ε, για να συζητήσουμε το θέμα και κυρίως την τρέχουσα κατάσταση για το ICS και τα καλά νέα είναι ότι μας ανέφεραν ότι η συμφωνία έχει συναυθεί. Επιβεβαιωθήκε και με μια συζήτηση εδώ χθε και όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουμε το κείμενο ICS είναι ε, ε, το ΣΥΤΑ ε, το οποίο είναι επίσης καλά νέο. Η συμφωνία φαίνεται ότι θα χωριστεί. Θα υπάρξει μια συνάντηση στην ομάδα παρακολούθησης. Έγινε η συζήτηση και εδώ χθε. Θα χωριστεί λοιπόν και θα μας το στείλουν τον Ιανουάριο και θα προχωρήσουμε στην επικύρωση. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις προς οποιονδήποτε από τους ηγητέ. Όχι. Οπότε κλείνουμε το σημείο αυτό και πάμε στο 21. Κανόνες και γενικές αρχές ε, σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη-μέλη της άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Και δίνω το λόγο στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Βαντεκάμπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Το ζήτημα αυτό είναι τεχνικό, περίπλοκο, αφορά την επιτροπολογία. και την ε, ε, πιο γρήγορη εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων. Μέχρι σήμερα ελάχιστη είναι η βούληση των κρατών μελών να συνεργαστούν ε, με τον απαραίτητο ρυθμό και η Κομισιόν έχει κάνει τέσσερις προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης ειδικότερα όσον αφορά τη συμπερίληψη των διαφορών μελών της ε, ε, ειδικής πλειοψηφία. να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο και πρόεδρε για να γνωστοποιείται το, η έκβαση των ψηφοφοριών στον κόσμο να γνωρίζει τι συμβαίνει. Είναι ένα πολύ τεχνικό ζήτημα. Ε, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας. Ε, γι' αυτό το λόγο έχω υποβάλει την τροπολογία 6α, όπου προτείνω η διαδικασία της Επιτροπής να μην οδηγούν σε καθυστέρηση των TDI. Επίσης αυτό το ε, θέμα να μην ε, παρέμβει στο, να μην επηρεάσει τον εξυγχρονισμό των TDI για το οποίο είναι η ο κ. Τσόνα. Αυτά είχα να πω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα στους κοιότης. Ο κύριος Μοέλ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια έκθεση πράγματι πολύ τεχνική, αλλά γύρει πραγματικά πολιτικά ερωτήματα γιατί πρόκειται για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων. Είχαμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε, όμως η διαδικασία επιτροπολογίας έχει γύρει θυελώδεις συζητήσεις, αντιδράσεις, σφοδρές κριτικές και επικρίσεις, κυρίως στο παρελθόν, ε, και εγκαλούσε τους πολιτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Περιθωριακά μόνο η Επιτροπολογία αφορά στην εμπορική πολιτική, αλλά είχαμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο των φωτοβολταϊκών πάνελ από την Κίνα, μεταξύ άλλων. Επομένως πρέπει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες. Είμαι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν τα λύνει όλα τα ζητήματα, αλλά τουλάχιστον πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και συμμερίζομαι και τις ανησυχίες του εισηγητή. Στηρίζω τις προτάσεις του έτσι ώστε η λήψη των αποφάσεων να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σε ό,τι με αφορά θέλω να προσθέσω δύο-τρία πράγματα που ενδεχομένως θα πάρουν τη μορφή τροπολογίας για να περιορίσουμε τον αριθμό των των αποχών που θα δηλώνει ένα κράτος μέλος και στη διαδικασία προσφυγών, ενώπιον της Επιτροπής των Προσφυγών, τη δευτεροβάθμια δηλαδή διαδικασία, και όταν πρόκειται για την επανα, επανεισαγωγή των μέτρων κατά του ντάμπινγκ. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχει και το Κοινοβούλιο περισσότερο δικαίωμα επίβλεψης ε, στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Εξόψεως είναι τεχνικό το ζήτημα κύριε Πρόεδρε, αλλά στην ουσία του είναι βαθύτατα πολιτικό. γιατί την ο κύριος Σόλτς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Φαίνεται να είναι τεχνική έκθεση και μάλιστα και αρκετά περίπλοκη. Αν το συγκρίνουμε όμως αυτό το θέμα με τη χθεσινή συζήτηση για τα ευρήματα του ελεκτικού συνεδρίου, τότε αντιλαμβανόμαστε πλήρως πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επομένως, επί της αρχής συμφωνούμε με την πρόταση γιατί κομίζει περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει να αναλυθεί πως αυτό το νέο σύστημα ακόμα και σε επίπεδο επιτροπών θεσπίζει αλλαγές στο πώς θα δηλώνονται οι αποχές εντός Συμβουλίου σε αυτή το περίπλοκο σύστημα καταμέτρησης των ψήφων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, οι εποχές καταμετρώνται, προσμετρώνται ως κατάστα σύστημα της ειδική πλειοψηφίας. Όμως κανονικά δεν μπαίνουν στη ψηφοφορία και δεν μπορούν να προσμετρηθούν ως κατά και γι' αυτό εμείς δεν είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ε, τις ψήφους αποχών δεν θα τις υπολογίζει στις ψήφους των παρόντων για την καταμέτρηση. Ε, με επιφύλαξη αντιμετωπίζουμε τη σύντμηση και συντόμευση των χρονικών περιθωρίων, γιατί μειώνεται έτσι ο ρόλος και η δυνατότητα να ασκήσει το ρόλο του το δημοκρατικό σώμα που έχει πλήρη νομιμοποίηση βεβαίως πρέπει να διατηρήσουμε την ικανότητά μας να έχουμε διαφάνεια και έλεγχο ταυτόχρονα. Από εκεί και πέρα, μια γενική παρατήρηση για τις εφαρμοστικές πράξεις. Το, μόνο το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα εξέτασης των ε, εφαρμοστικών πράξεων και παρόλο που δεν είναι αυτός ο στόχος της επιστολής προτάσεων αυτής, πρέπει να ζητήσουμε να ενισχυθούν οι δικές μας εξουσίες και αρμοδιότητες γιατί είμαστε νομοθέτες. Θα μπορούσε να προτείνει το Κοινοβούλιο και να παρουσιάσει γνωμοδότηση ή τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα της άρνηση κυρίας για τις εφαρμοστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Ο κύριος Μπούχνερ δεν θέλει το λόγο για τους πρασίνους, οπότε η Επιτροπή. Ο κύριος Χένινγκ και η κυρία Γιαμπόα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ήδη συζητήσει με τον εισηγητή στις 30 Αυγούστου για το θέμα αυτό. Να υπενθυμίσω. τι προσπαθεί να επιλύσει η Κομισιόν. Ένα πολύ περιορισμένο και συγκεκριμένο πρόβλημα. Ε, θεωρούμε ότι η επιτροπολογία και το υπάρχον πλαίσιο λειτουργούν πολύ καλά και θα μπορούσα να το τεκμηριώσω με ένα μόνο στοιχείο. Έχουμε κάθε χρόνο γύρω στις 1500 εκτελεστικές πράξεις. μόνο μία ή δύο καταλήγουν σε κατάσταση καμία άποψη που σημαίνει πως δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά. Το 2015 για παράδειγμα είχαμε 1700 ε, εκτελεστικές πράξεις. Οι 36 κατέληξαν σε καμία άποψη και μόνο 15 από αυτέ τι 36 χρειάστηκε να περάσουν στην Επιτροπή Πανεξέτασης. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα, γιατί αυτές οι 15 είναι μεν πολύ λίγε, αλλά αφορούσαν πολύ ευαίσθητα θέματα. Αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Κομισιόν σε τελευταία ανάλυση. Η Κομισιόν πρέπει να πάρει μια απόφαση. Αν δεν υπάρχει σαφής άποψη μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κατέληξαν σε σαφή άποψη δεν ήταν διατεθειμένα να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες παρά ότι σε τελευταία ανάλυση ως νομοθέτες παρέχουν ε, τη νομική βάση, το νομικό πλαίσιο. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Επιτροπή και γι' αυτό προτείνουμε να αλλάξουν οι κανόνες για την ψηφοφορία, ώστε να έχουν κίνητρα οι χώρες να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία. Να πω κάτι για τις τροπολογίες του εισηγητή. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που αφορούν τις προθεσμίες ε, στον τομέα του εμπορίου και τα αντίμετρα. Δεν νομίζουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, προκαλούν προβλήματα. Για παράδειγμα, η δεύτερη αναπομπή στην Επιτροπή Επανεξέτασης ή Εφέσεων είναι μόνο μια δυνατότητα, δεν υποχρεωτική. Και αν υπάρξει αναπομπή στο Συμβούλιο για μια άτυπη συζήτηση, υπάρχει δυνατότητα να περικοπεί η προθεσμία. Ο εισηγητής προτείνει να υπάρξει ε, περίοδος χάριτος ε, ενός μήνα μεταξύ της έγκρισης από την Επιτροπή και της εξέτασης στο Συμβούλιο υπήρχε στον κανονισμό αλλά κάποια στιγμή καταργήθηκε γιατί είχε οδηγήσει σε κάποιες ακαμψίες στην πραγματικότητα η περίοδος μεταξύ της εξέτασης από την προπολογία και της τελικής έγκρισης από την Επιτροπή της εκτελεστικη πραξης πράξης είναι 30-40 μέρε. Οπότε μπορούμε να έχουμε μια περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μάλλον όχι. Ε, προτιμούμε να μην υπάρξει περίοδο λοιπόν του ενό μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα σχόλια του, σκιώδου από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ για το σχόλιο της Γκουε. Έτσι η πολιτική συζήτηση για τι τροπολογίε θα ζωηρέψει λίγο. Με ενδιαφέρουν όλα τα σημεία τα οποία ακούσαμε ε, στα σχόλια ε, και όπως ε, πάντα θα λάβουμε υπόψη και τα σχόλια της Κομισιόν. Δεν θέλω να λάβω κάποια θέση αυτή τη στιγμή, αλλά θα συζητήσω με τους Κιώδης για τη θέση της Κομισιόν και θα καταλήξω όπως γνωρίζετε σε μια ε, σοφή θέση και απόφαση. Μα και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει σοφή απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τελειώσαμε με το 21. Προθεσμία για τις τροπολογίες 20 Οκτωβρίου, 12 η ώρα. 20 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο Χέρμουντ Σόλτ πρέπει να μας στείλει τις τροπολογίες του. Άριστα. Περνάμε στο 22. περαιτέρω ανάπτυξη, επέκταση των κεφαλαίων για, την, για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες. Έχουμε την παράδοση. Οι πιο πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες να περιέχουν ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη το 2011 στη συμφωνία με την Κορέα υπήρχε ένα εκτεταμένο κεφάλαιο για το θέμα αυτό και έχει αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η διάσταση των εμπορικών ε, συμφωνιών. Τους τελευταίους μήνες ιδιαίτερα στα πλαίσια της συζήτησης για το TTIP και για τη συμφωνία με τον Καναδά. Τη ΣΕΤΑ δηλαδή. Αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο αυτό το κεφάλαιο εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε τίθεται το ερώτημα. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και τίθεται ιδιαίτερα τρία θέματα. Και γι' αυτό το θέσαμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο. Εάν θέλουμε να υπάρξει περαιτέρω εδραίωση του κεφαλαίου αυτού και περαιτέρω διαστάσεις να συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό. Για παράδειγμα, αυτό που είχε προταθεί για το TTIP είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Ποιοτικά, πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε διαρωτώ με. Πώς είναι δυνατόν στις διαπραγματεύσεις που έχουμε τώρα για παράδειγμα με το Μεξικό ή με το Μερκοσούρ να το κεφάλαιο για το θέμα αυτό, Το οποίο υπολείπονται πολύ τη κατάσταση του TTIP. Δηλαδή η σημειωθήσα πρόοδο μοιάζει να έχει ε, αντιστραφεί. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα το ενέκρινε αυτό. Μας υποβάλλονται συμφωνίες που υπολείπονται πολύ των αντιστοίχων κεφαλαίων της ΣΕΤΑ. Πώς είναι δυνατόν να μας υποβάλουν... Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο ζήτημα, στη δεύτερο σημείο. Έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω αυτές ε, τις εξελίξεις και ότι θέλουμε στις, και συμφωνήσαμε ρητά στη ΣΕΤΑ να αξιοποιήσουμε πλήρως ε, ε, τη συμφωνία αυτή με μια περαιτέρω εξέλιξη, με μια επιβολή του κεφαλαίου εμπορίου και βιωσιμότητας. Στις 21 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε πλήρη η ΣΕΤΑ και δεν έχω μάθει ε, πώς αυτή η διαδικασία της επιβολής ε, πρόκειται να εξελιχθεί. Υπάρχουν κάποια κενά. Οπότε είναι αναγκαίο να συζητήσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για τη διαδικασία επιβολής. Ε, που συμφωνήθηκε κατά τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Και αυτό με φέρει στο τρίτο μου σημείο. Ε, υπάρχει ένα non-paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ουσιαστικά δεν ξέρω το non-paper είναι μια επίσημη δήλωση της Κομισιόν υπάρχει, κρύβεται κάτι από πίσω τι χαρακτήρα έχει ακριβώς ένα non-paper είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Παρ' όλα αυτά, εκεί μέσα διαπιστώνει κανείς ότι κατά βάση δύο επιλογές περιγράφονται. Η πρώτη, προχωράμε όπως έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και η δεύτερη, ε, παίρνουμε το μοντέλο των ΙΠΑ. Εάν ακολουθήσουμε το μοντέλο των ΗΠΑ, αυτό εδώ στο ε, Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να υποστηριχθεί. Ε, το είχαμε συζητήσει με τη Γουατεμάλα. Και ε, είχαμε πει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδειχθεί ε, ότι έχει αποτελέσματα. και επίση ε, συμπεριλάμβανε η όλη διαδικασία κυρώσεις ε, φαίνονταν καλή διαδικασία αλλά υπάρχει μια σειρά συζητήσεων όπου εναλλασσόμαστε μεταξύ ε, μαύρου και άσπρου ε, και εγώ είχα κάνει και μια πρόταση να πάρουμε τα θετικά της ευρωπαϊκής προσέγγισης, το διάλογο, το πάνελ εμπειρογνωμόνων ως αρχή ε, λήψης αποφάσεων και να έχουμε και ένα μηχανισμό επιβολής ο οποίος θα οδηγήσει ε, το πάνελ των εμπειρογνωμόνων να οδηγήσει σε ε, υποχρεωτικούς μηχανισμούς και σε αποζημιώσεις ουσιαστικά, σε αντιστάθμιση. για να μπορούν να λαμβάνουν αποζημιώσεις ε, για τις ε, ζημίες που θα έχουν υποστεί τα συνδικάτα και εργαζόμενοι. Και όλα αυτά δεν είναι μέσα σε αυτό το non-paper. Θέτω λοιπόν αυτά τα τρία θέματα. Και ρωτώ ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά λόγω του ότι ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς είχε ήδη το Μάιο πει ότι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων. Επ' αυτού δεν βλέπω καμία πρόοδο μέχρι στιγμής. Αυτά ως εισαγωγή. Και τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτη η Τζουντ. Κύριε Ντάρλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι αξίζεται εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο έχετε προχωρήσει αυτό το πολιτικό πρόγραμμα, τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλετε προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφέστατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται έμπνευση και οι προτάσεις που υποβάλλετε που έχουν υποβληθεί είναι απαξιωμένες και έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και πολύ σωστά το είπατε εσείς αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα και να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει παντού στον κόσμο. Ο σχετικός δείκτης δείχνει ότι ο αριθμός των χωρών όπου εργαζόμενοι υφίστανται σωματική βία και απειλές έχει αυξηθεί κατά 10% και πολλές χώρες που έχουν μπει μέσα στις 10 πρώτες σε αυτό το κατάλογο είναι χώρες με τις οποίες η, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνία ελεύθερων εμπορίου, ε, ελεύθερο ελεύθερων συναλλαγών και έχει και, και κεφάλαια σχετικά με την αηφόρο ανάπτυξη και το καθεξής. Τα στοιχεία λοιπόν είναι συντριπτικά για το πόσο καλά ή κακά, αν θέλετε, λειτουργεί αυτό το σύστημα το σημερινό του business as usual και του δεν τρέχει τίποτα. Ποια στοιχεία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την Κανά λέει ότι το δικό της μοντέλο είναι το αποτελεσματικό, το υφεστάμενο μοντέλο λειτουργεί. Και αν προτείνει αυτή η, αυτή προσέγγιση να υιοθετηθεί και στο μέλλον για το, ε, ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη, πώς το, ε, Πώς το στοιχειοθετεί αυτό. Η Νότια Κορέα έχει μόλις μπει στις 10 πρώτες χώρες στο κατάλογο του στο δίκτυο το σχετικό. Και βλέπουμε διάφορες ελλείψεις και ανεπάρκειες ε, σε θέματα εφόρου ανάπτυξης. Η διερευνητική αποστολή στην Νότιο Κορέα το κατέδειξε αυτό, το απέδειξε. Μία παραβίαση, για παράδειγμα, είναι η καταστολή των ε, συνδικάτων των καθηγητών και δασκάλων. Άλλο παράδειγμα είναι η Γουατεμάλα εκεί ως εμπορική πολιτική έχουμε φύγει από το GSP Sin, GSP Plus, σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν που, και τους περιορισμούς του που δεν εφαρμόζονται σωστά όταν έχουμε παραβιάσεις των κανόνων παραβάσεις των κανόνων και έχουμε πάει προς μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια όμως αυτό είναι πιο αδύναμο σε σχέση με το μοντέλο της Νοτιού Κορέας σε ό,τι αφορά την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και τις ανησυχίες και πόσο αυτές αναδεικνύονται. Ε, έχει χάσει την αξιοπιστία της αυτή η συμφωνία με την ε, Γουατεμάλα. Αν πρέπει κανείς να αποδείξει ότι η χή καταστρατήγηση του εργασιακής νομοθεσίας έχει πολύ συγκεκριμένη και απτή επίπτωση στο εμπόριο και αν δεν υπάρχει αυτή η απόδειξη να μην μπορεί να επικαλεστεί η καταστρατήγηση της συμφωνίας για να δράσει, ε, τότε ποτέ δεν θα αναλυφθεί καμία δράση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί αυτό με τον τρόπο τον τυπολατρικό που ε, προβάλλεται. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μπορεί να υπάρχει μία διαδικασία υποβολής προσφυγών, τα συνδικάτα να υποβάλουν προσφυγές για καταστρατήγηση του εργατικού δικαίου σε ανεξάρτητες αρχές, σε μια ομάδα συμβουλευτική, σε μια γραμματεία που θα μεριμνά και θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και θα μπορούσαν να γίνουν ανεξάρτητες έρευνες για αυτή την προσφυγή. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με τρόπο πολύ παρόμοιο με αυτόν που παρουσιάζεται στις δικές σας προτάσεις, κύριε Πρόεδρε. Να πάρουμε τα ενία να είμαστε διαφανείς, να έχουμε ανοιχτό πνεύμα και να ξεκαθαρίσουμε ποια κριτήρια ισχύουν και μάλιστα σε όλους τους συμμετέχοντες. Από εκεί και πέρα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθείται μια ήπια διπλωματική προσέγγιση, δεν αρκεί, είναι χρήσιμο το καρότο, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και μαστίγιο για να φάει ο γάιδαρος το καρότο ή κάποιο άλλο ζώο ή ίσως ε, το ανθρώπινο είδος, δεν εννοώ τίποτα άσχημο με αυτό. Ε, χρειαζόμαστε δηλαδή υλικέ και συγκεκριμένες κυρώσεις έτσι ώστε οι εταιρείε να αναλάβουν δράση και να διασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουν δράση μετά από προσφυγέ γιατί θα έχουν καταστρατηγήσει συγκεκριμένε ρήτρε τη συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Ήδη αλλιώ θα έχουμε πάλι την πολύ όμορφη πολυλογία που μα διακρίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα υψηλά πρότυπα τα εργασιακά χωρίς να κάνουμε τίποτα στην πράξη τα εργασιακά δίκαιο το εργασιακό δίκαιο και η περιβαλλοντική προστασία δεν θα πρέπει να μπαίνουν μόνο στο κεφάλαιο για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες και να μην περικλείονται και περιοριστικά να βρίσκονται μόνο εκεί αλλά και στα υπόλοιπα κεφάλαια της συμφωνίας. Θέλω να διευρύνω λίγο το βλέμμα, όχι μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε πολλές συμβάσεις, συμφωνίες, εμπλέγονται ορισμένα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αγνοούνται κατόπιν. Έχω την εντύπωση ότι κυρίως ε, ενδιαφέρει την Κομισιόν να αναπτύσσεται το εμπόριο, να κινείται το χρήμα, αλλά όχι ιδιαίτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να ασκήσουμε πολύ περισσότερη πίεση από ό,τι μέχρι στιγμής για να γίνουν πολύ πιο αξιόπιστα αυτά που λέγονται και όταν υπάρχουν παραβιάσεις να ελέγχονται. Δεν έχουμε κάνει ακόμη τη συζήτηση για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί για υποβολή παραπώνων, σημεία επαφής, με όνομα, διεύθυνση, email, ούτως ώστε τα θύματα να μπορούν να αποζημιώνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βίνκλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εμείς διαβάσαμε αυτό το non-paper από την Κομισιόν που δεν σας αρέσει σας από ό,τι φαίνεται και συζητάμε εντός του ΕΛΚ πώς να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία των εμπορικών συμφωνιών ε, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των νέων κεφαλαίων. Όταν αποφάσισε η Ένωση να συμπεριληφθούν τέτοια κεφάλαια σε αυτές τις συμφωνίες, το έκανε γιατί είχε συνείδηση του ότι πρέπει να προωθήσουμε τις αρχές μας. Τα κεφάλαια αυτά, αν τα εξετάσουμε, έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής και ενισχύουν το πολυμερές σύστημα. Και φυσικά πρέπει να συμβάλλουν στην καλή διακυβέρνηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όπως ήδη υπόθηκε και τονίστηκε Άρα πρέπει να συνεργαστούμε με τους διεθνείς οργανισμούς, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας πρώτα απ' όλα. Πρέπει να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία. Επίσης έχουμε τους οργανισμούς που δημιουργούνται μέσω των ε, διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλη τη γνώση που υπάρχει. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε καλύτερα με τους εμπορικούς μας εταίρους. Και όπως και εσείς αναφέρατε, Πρόεδρε, πρέπει να εφαρμοστούν ήδη τα ισχύοντα κεφάλαια, κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς επιτηρούμε την εφαρμογή αυτών των κεφαλαίων. Έχουν δεσμευθεί οι εταίροι μας, αλλά τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Πλήρως. Υπάρχει ένας μηχανισμός για την επίλυση διαφορών για την εφαρμογή αυτών των κεφαλαίων, αλλά δεν ξέρω αν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτοί οι μηχανισμοί. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε τους υπάρχοντες μηχανισμούς πριν αρχίσουμε να συζητάμε τη δημιουργία άλλων κατά τη γνώμη του ΕΛΚ. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε τι γίνεται επί τόπου, πώς λειτουργούν οι τοπικοί μηχανισμοί εποπτείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει επί τόπου. Γίνονται όσα πρέπει να γίνονται. Η πραγματικότητα επί τόπου είναι αυτή που νομίζουμε ή και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης γιατί έχουμε αντιπροσωπείες της Ένωσης ε, στις χώρες αυτές. Έχουμε πρεσβείες των κρατών μελών. Έχουμε τα ενωσιακά εμπορικά επιμελητήρια. Αξιοποιούμε όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες για να εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί, για να προωθούνται οι αξίες μας. Αυτά είναι τα θέματα θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε και να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Τώρα που ε, πλησιάζει και η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της στρατηγικής μας για τα θέματα αυτά. Οπότε αυτή η μεσοπρόθεσμη επανεξέταση είναι κατάλληλη ευκαιρία για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Πρόεδρος, ναι βεβαίως, λέει ο πρόεδρος, ναι είναι τμήμα της συζήτησης εμπόριο για όλους. Τον Νοέμβριο θα έχουμε και την ημερίδα για την εμπορική πολιτική. Ο Χέλμουντ Σόλτ. Ευχαριστώ. Να εξετάσω πρώτα απ' όλα μία άλλη άποψη. Κατά τη συζήτηση δεν έχουμε εδώ συναδέλφους από το Άλντε και το ΕΛΚ που ήταν εδώ παρόντες για τις εμπορικές συμφωνίες και μάλιστα απέρριψαν τις τροπολογίες άγκρι που κυρίως προσπαθούσαν να προωθήσουν τα συμφέροντα των τοπικών παραγωγών, ε, την προστασία του περιβάλλοντος. Όταν σήμερα συζητάμε για την υπεύθυνη στάση που πρέπει να έχουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα αυτό σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη. Θέλω να πω συγκεκριμένα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προσέγγιση της εμπόριο για όλους, προσπάθησε να προωθεί στα θέματα αυτά και μετά από πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινή γνώμης. Και αυτή η νέα προσέγγιση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από το Global Europe. Και βεβαίως ε, συμφωνώ με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν, που είπαν πώς πραγματικά θα καταλήξουμε σε μηχανισμούς πραγματικής επιτήρησης της εφαρμογής Συμφωνώ. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε όλοι. Αλλά τι γίνεται μετά στις ψηφοφορίες, εκεί προκύπτουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Άρα το θέμα είναι με πόση σοβαρότητα εφαρμόζουμε αυτά τα οποία αποφασίζουμε. Χθες ε, συζητήσαμε τα θέματα της οικονομίας σε σχέση με το εμπόριο και είπαμε ποιος αποφασίζει τους κανόνες. Τι ρόλο παίζουν αυτά τα κεφάλαια. Πώς επηρεάζουν την ε, κατάσταση επιτόπου. Πώς επηρεάζουμε τις αλυσίδες παραγωγής. Γιατί ξέρουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα του εμπορίου γίνεται εντός των πολυεθνικών ομίλων, όπου δεν μπορεί να παρεύει το κράτος. Τι κάνουμε εκεί, προσπαθούμε να μπούμε εκεί πέρα μέσα, να βάλουμε το κεφάλαιο με βιώσιμες ανάδειξεις και σε αυτές τις συναλλαγές. Γιατί είναι μια δυνατότητα. να τροποποιήσουμε τις παγκόσμιες διαδικασίες δημιουργίας αξίας προς το συμφέρον του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εργαζομένων, να τα αναδιαμορφώσουμε όλα αυτά, να τα βελτιώσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας και ιδιαίτερα εμείς στο Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι βεβαίως, βεβαίω, σωστό ότι η Επιτροπή χρειάζεται τη δική μας πίεση και στήριξη για να τα προωθεί στα θέματα αυτά. Και τώρα, σύντομα ορισμένα άλλα. Για τις εργασιακές ε, προδιαγραφές, αν δούμε τι γίνεται στη συμφωνία με το Μεξικό. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην ε, προδιαγραφή του 98 για τους ε, κοινωνικούς εταίρους γίνεται αναφορά μόνο στις ε, διατάξεις του 1969. Εμάς μας ενδιαφέρει και η προστασία των ε, κοινοτήτων των αυτοχθόνων, όπως είπε και ο Κλάους Μπούχνερ. Υπάρχουν παραδοσιακά ε, εργασιακά δικαιώματα, δικαιώματα εργαζομένων, αλλά και τα ευρύτερα ανθρώπινα δικαιώματα για το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γιατί δεν γίνεται αναφορά στα εθνικά σχέδια εφαρμογής. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ε, ε, είναι περίπλοκη η σύνδεση των εθνικών με τους διεθνείς στόχους και σχέδια. Και συμφωνώ με τον κύριο Βίνκλερ. Σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να δούμε γιατί μέχρι στιγμής δεν λειτουργούν οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, οι μηχανισμοί διατησίας. Και αυτό είναι το τμήμα της συζήτησης. Επίσης, υπάρχει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Συνδικάτων. Είναι αναλυτικό έγγραφο, περιέχει διάφορες προτάσεις, πολλά στοιχεία για τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια αυτών των κεφαλαίων ανεξάρτητα από τις δύο εναλλακτικέ που περιέχει αυτό το non-paper Ούτω ώστε να ενισχύσουμε αυτά τα κεφάλαια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Είμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θέλω να σας επισημάνω το γεγονός ότι παρεμβαίνω εξ ονόματος της κυρίας Αλέσια Μόσα για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η οποία χρειάστηκε να πάει στην εκλογική της περιφέρεια. Και μετά θα σας πω τη δική μου άποψη. Καλωσορίζουμε το non-paper για το εμπόριο και την αηφοροανάπτυξη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι. Εκτιμούμε την ειλικρίνεια με την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει τα προβλήματα του υφιστάμενου καθεστώτος και δεσμεύεται να κάνει συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επομένως, με έκπληξη ανακαλύψαμε ότι η πρόταση για τα κεφάλαια για το εμπόριο και η φόρα ανάπτυξη στις διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ και το Μεξικό στη πράξη μοιάζουν πάρα πολύ με τις ήδη ισχύουσε ε, συμφωνίες και συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας εξετάσει το, τη πολύ μικρή χρονική πρεθεσμία για τις δύο αυτές συμφωνίες ή συμβάσεις. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το ότι η Επιτροπή προτείνει κάτι με το οποίο δεν είναι ικανοποιημένη ούτε η ίδια και το οποίο βεβαίως δεν ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά τις, ε, το οικονομικό όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Νότιο ε, Κορέα κατέδειξε πόσο αδύναμες είναι οι διατάξεις αυτές για το εμπόριο και την αηφόρο ανάπτυξη. Έχει υπάρξει δέσμευση για μηχανισμό αναθεώρησης έτσι ώστε τα σχετικά κεφάλαια να μπορούν να τεθούν σε ισχύ και να εφαρμόζονται. Μια νέα συμφωνία πρέπει να χτιστεί πάνω στο κεκτημένο της ΣΕΤΑ. Επομένως είναι απαράδεκτο η Συμφωνία ΕΕ Ιαπωνία να μην περιλαμβάνει αυτό το μηχανισμό αναθεώρησης ή επανεξέτασης. Θα θέλαμε να ξέραμε λοιπόν το γιατί. Έχοντας ε, κηρύξει την έναρξη της συζήτησης της σχετικής, γιατί μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι προτάσεις για τη Μερκοσούρ και το Μεξικό δεν θα περιλαμβάνουν τίποτα για την ειδική υποχρέωση των μερών να προωθήσουν τη συμμόρφωση και να θέσουν σε ισχύ του το χώριο περιβαλλοντικό και εργατικό δίκαιο. Όταν μιλούμε για μηχανισμό που θα βασίζεται σε κυρώσεις, οι σοσιαλιστές δεν θέλουν αυτός να αντικαταστήσει τα εργαλεία συνεργασίας και διαλόγου. Αντιθέτως, το θέλουμε ως τελευταία προσφυγή. Ε, ένα μηχανισμό που θα αυξήσει το κινητήριο, θα εντείνει το κινητήριο μοχλό που έχουμε για να ε, παρακινήσουμε τους εταίρους μας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις μας, τους. Αυτή είναι η παρέμβαση της συντονίστριας και τώρα θέλω να εκφράσω την προσωπική μου άποψη παρακαλώ. Έχω λοιπόν μια ερώτηση που θέλω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, ως προς τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που, δε, που ισχύουν ήδη και δεν έχουν κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη γιατί όταν συνήφθησαν αυτές οι συμφωνίες δεν γινόταν λόγος για κάτι τέτοιο περιπτώσει. Για αυτές τις συμφωνίες λοιπόν έχετε σκεφτεί ως Επιτροπή να υπάρξει κάποιος μηχανισμός που θα επιτρέπει ε, να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να χρειάζεται να ξαναξεκινήσουμε την επανεξέταση και αναθεώρηση του συνόλου της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνίες με διαφορετικές προϋποθέσεις και διαφορετικές συνθήκες με, τη, με τις διάφορες χώρες. Ε, τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά απαιτούν να έχουμε κεφάλαιο για τα ζητήματα αυτά, τα οποία υπάρχουν παντού. Υπενθυμίζω την ανάγκη να υπάρχει ένας τρόπος να εκτελείται, να εφαρμόζεται στην πραγματικότητα το σχετικό κεφάλαιο. Και αναφέρομαι βεβαίως στη συμφωνία με την Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων. Και τέλος, ένας μηχανισμός που θα βασίζεται σε κυρώσεις. Υπ' αυτή την έννοια, δεν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταυρώνει τα χέρια μπροστά σε ένα αίτημα που είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία. Με το ISTS το είδαμε να συμβαίνει για άλλη μια φορά. Οι οργανώσεις πολιτών, οι κοινωνικές οργανώσεις, πολιτικές ομάδες άσκησαν πολύ μεγάλη πίεση και η δική μου πολιτική ομάδα βεβαίως και στη συνέχεια όταν αναθεωρηθεί και το σύστημα και ε, παρετηθήκαμε από το σύστημα ιδιωτικής διαιτησίας. Θυμάμαι ε, προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ίδια την Επίτροπο να λέει ότι δεν μπορεί να ξανανοίξει η Συμφωνία ΣΕΤΑ. Εμείς αυτό απαντήσαμε ότι δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια συμφωνία που να περιλαμβάνουν ε, αυτά τα ζητήματα και μετά ξανά άνοιξαν διαπραγματεύσεις όταν είπαμε ότι δεν θα το ψηφίζαμε και βρέθηκε τρόπος. Άρα είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η συζήτηση για το ποιο είναι το καλύτερο σύστημα, για το ποιο είναι ένας μηχανισμός που θα βασίζεται σε κυρώσεις, που θα λειτουργεί αποτρεπτικά, αποτρεπτικά προς ε, χώρες που έχουν συστήματα που πλήττουν τις αξίες και τις αρχές μας. Και θέλω να παρουσιάσω και ένα παράδειγμα, Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω. Είχαμε ένα δίκτυο ε, τρομακτικής σοβαρότητας των οδικών ατυχημάτων. Και επειδή οι κυρώσεις και τα πρόστιμα δεν, ήταν, δεν έφταναν, βάλαμε ένα point system. Κάθε οδηγός μάζευε πόντους και όσο περισσότερες οδικές παραβάσεις είχε διάφορους πόντους και με τις παραβάσεις του αφαιρούνται πόντι μέχρι ότου να του αφαιρεθεί και η άδεια οδήγηση στο δίπλωμα. Και τελικά μειώθηκαν τα ποσοστά ε, κατά 50% με αυτό το point system. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Τιτσιάνα Μπέγγιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ του να συμπεριλάβουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα σχετικά κεφάλαια στη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Το λέω σε κάθε ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταλάβει και συμπεριλάβει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη όλες τις συμφωνίες. Καμιά φορά με διαφορετικές διατάξεις, αλλά παντού με κάτι κοινό. Κάτι που επαναλαμβάνω εγώ διαρκώ όταν αναφέρομαι σε αυτά τα κεφάλαια. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικέ κυρώσει. Όπω λένε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν ξέρουμε αν η παραβίαση των υποχρέωσεων της βιώσιμης ανάπτυξε μια ε, συμφωνία μπορεί να διωχθεί μέσω κάποιου μηχανισμού επίλυσης διαφορών ε, μεταξύ κρατών. Αλλά και να υπάρχει τέτοια κύρωση ε, αμφιβάλλω κατά πόσο θα ε, δει κάποιο κράτος ένα Ένα άλλο. Γι' αυτό το λόγο είναι απολύτω απαραίτητη η συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, ώστε οι κυρώσει να λειτουργούν πραγματικά. Γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα τι αναλυτικέ Προτάσει της ε, μελέτης ε, που ανέθεσε ο πρόεδρος κ. Λάγκε πιο φιλόδοξες προτάσει από αυτές τις Κομισιόν. Αλλά από ό,τι κατάλαβα η Κομισιόν διάλεξε άλλη οδό. Για παράδειγμα στη συμφωνία με το Βιετνάμ δεν προβλέπονται κυρώσεις και αυτή η επιλογή είναι περίεργη. Ε, κυρίως επειδή το Βιετνάμ είχε συμφωνήσει να υπάρχουν κυρώσεις στην Συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ. Οπότε ρωτάω την Κομισιόν γιατί κάνατε αυτή την επιλογή με ε, τον εταίρο μας αυτό στην Ασία. Τέλος, θα ήθελα να δω μια πραγματική δέσμευση των διαπραγματευτών για τα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης. Αναμφίβολα θα συνέβαλε σημαντικά στην νομιμοποίηση της εμπορικής πολιτικής και στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, ε, οργανισμού που προωθεί τα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Άλμα ε, Μένιερ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Μινέρ. Έχω δύο ακόμες παρατηρήσεις ε, που μπορεί να σχετίζονται με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Θα ήθελα να υπήρχαν και περισσότεροι εδώ. Είναι κρίμα που θεωρούν κάποιοι ότι αυτά που, που λέμε εμείς από την πλευρά μας δεν είναι σημαντικά. Τον Ιούλιο εμφανίστηκε ένα νέο non-paper της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εμπορικοί εταίροι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριέλαβαν τις περιβαλλοντικές πτυχές ε, ε, εδώ και μερικά χρόνια. Υπάρχουν δεσμευτικοί μηχανισμοί, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Πώς είναι λοιπόν δεσμευτικοί. Πώς είναι δεσμευτικά τέτοια μέτρα. Δύο επιλογές παρέχονται στο έγγραφο. Η μία είναι κάποιο είδου εταιρική σχέση με χώρε εταίρου και η δεύτερη είναι μια επιλογή με κυρώσει. Και η Κομισιόν χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό με τη Γουατεμάλα μέσω του οποίου προσπαθεί να αμφισβητήσει αυτά τα μοντέλα, να πει ότι δεν λειτουργούν, αλλά αυτό δεν αληθεύει. αυτό έχει καταστρέφει και σε κάποιο ε, αντίδραση που έχει συνταχθεί από κάποιον για αυτό το θέμα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Κομισιόν δεν φέρνει καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε ε, στη συμφωνία με την Νότια Κορέα. Παρατηρούμε ότι χρόνια διπλωματικών προσπαθειών δεν ε, έχουν αλλάξει τίποτα. Ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται υπό απάνθρωπες συνθήκες παρά όλες αυτές τις συνομιλίες. Αν δούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στι συμφωνίε με το Μεξικό και με τι χώρε Μερκοσούρ, υπάρχουν πολλά κενά. Στο Μεξικό δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά την εμπορία ε, ειδών τη και την παρανομιλοτομία και στη συμφωνία με τι χώρε Μερκοσούρ η συμφωνία του ILO δεν έχει επικυρωθεί ενώ θα έπρεπε να αποτελεί προαπαιτούμενο κατά την απόψή μας. Επίσης ε, αναφέρουμε τις βεβαιώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις συμφωνίες. Θα πρέπει αυτές οι διατάξεις να συνεπάγονται κυρώσεις, ε, συνέπειες. Επίσης θα υποστηρίζαμε ε, να υπάρχει κάτι δεσμευτικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πέραν αυτού δεν πρέπει να ξεχνάμε τις προτεραιότητες που έχουμε δώσει σε διάφορες συμφωνίες του ΠΟΕ και λοιπές όπως φαίνεται δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην βιωσιμότητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη βιωσιμότητα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ και η Καρολίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια συνεδρίαση των συντονιστών για την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία κατά την οποία συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Κομισιόν ότι πρέπει τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη να είναι ισχυρά στις συμφωνίες. Αλλά δεν συμφωνήσαμε τελικά τι ακριβώς θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτό μας το μήνυμα η οικονομική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να γίνεται όμως πιστεύω σε βάρος του περιβάλλοντος ή των εργαζομένων. Αλλά τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη. Ναι, ναι, λέμε, α παρακαλούμε μην τα κάνετε αυτά και όταν δεν τα τηρούν δεν έχουμε καμία δυνατότητα να επιβάλλουμε την άποψή μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Όταν υπάρχουν παραβάσεις πρέπει να έχουμε δυνατότητα να αντιδράσουμε. Πρέπει να έχουν επιπτώσει οι ενεργειές τους. Συμφωνούμε. Χρειάζονται κυρώσει. Κάποιας μορφής. Ξέρω ότι ίσως δεν είναι στην αρχή η κατάλληλη στιγμή να διατυπώσουμε αυτέ τι απαιτήσει, γιατί ίσω να μην δημιουργήσει πνεύμα εμπιστοσύνη. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη έναντι των συμπολιτών μα. Να είναι πεπισμένοι, ναι, είναι καλέ οι εμπορικέ συμφωνίε, αλλά αν δεν εφαρμοστούν σωστά, τότε θα υπάρξουν αντιδράσει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κυρώσει. Δεσμευτικέ κυρώσει. Μόνο τότε είμαστε αξιόπιστοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη προ του εταίρου μα, αλλά όπω ένα γάμο. Είναι αν όλα είναι καλά, όλα είναι θαυμάσια, δεν χρειάζονται νόμοι αλλά όταν ε, θες να πάρεις διαζύγιο τότε χρειάζονται κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να είναι φιλόδοξη η προσέγγιση της Κομισιόν. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, οπωσδήποτε να συμμετέχει. Έτσι κερδίζουμε όλοι. Δεν αρκούν εθελούσιες διατάξεις. Δεν μπορούν έτσι να λειτουργήσουν συμφωνίες. Χρειάζονται κυρώσεις που θα εφαρμόζονται μόνο εάν χρειάζεται. Θα πρέπει να ελέγχουμε εάν εφαρμόζεται αυτό που αποφασίσαμε, γι' αυτό χρειάζονται αυτές οι ομάδες επίβλεψης για να δούμε πώς λειτουργεί η συμφωνία και τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν λειτουργεί. Πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα, να επιβάλλουμε τα κατάλληλα μέτρα και γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτός είναι ο στόχος μας θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν ε, στις σχέσεις με όλα τα κράτη, τις εμπορικές. Σε όλες τις ε, τέτοιες συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο να ισχύουν αυτές οι διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Μαντλέν. Λοιπόν, οι συζητήσεις μας νωρίτερα το πρωί ε, ήταν πιο αρμονικές, τώρα είναι λίγο πιο έντονες. Αλλά σας παρακαλώ να αντιδράσετε στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Η ομορφιά αυτής της συζήτησης έγκυται στο γεγονός ότι τελικά διαπιστώνει κανείς σύγκληση και φαίνεται βέβαια από την άλλη όταν φτάσουμε σε κάποια φλέγοντα ζητήματα ότι έχουμε δυνάμεις αποκλίνουσες. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς αντιλαμβάνεται κανείς το εφικτό και τι αντιλαμβάνεται κανείς ως εφικτό. Εγώ δεν νομίζω ότι φτάνουμε στη σύγκληση. Ακούω τις παρατηρήσεις σας και τις σημειώνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα non-paper, ένα έγγραφο συζήτησης δηλαδή που έστειλε στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη για να γίνει συζήτηση. Αυτό θέλουμε. Δεν υπάρχει κάποιο ε, κάποιος επίσημος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να απαντήσετε. Εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και θέλαμε να είναι όσο να τον πιο ε, ευρεία η λίστα των συμμετοχόντων. Τη βάλαμε στην ιστοσελίδα μας και από τον Ιούλιο είμαστε στο δρόμο. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό συναντήσεις στις Βρυξέλλες, ε, συναντήσεις ατομικά, ξεχωριστά με τα κράτη-μέλη, με ειδικού, με συνομιλητές και αύριο το ίδιο έχουμε πάει σε πέντε πρωτεύουσε για να συζητήσουμε με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και και στις Βρυξέλλες συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών και η ΕΤΟΚ με περιβαλλοντικές με κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες ε, βρίθουμε από συζητήσεις και από επικοινωνίες και επαφές. Χρειάστηκε χρόνος για να υπάρξουν αντιδράσεις, άρα συμπεραίνω ότι η συζήτηση δεν είναι εύκολη. Πολλοί συντάσσουν έγγραφα που θέλουν να μας στείλουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να δώσουμε χρόνο για να υπάρξουν αυτά και να μην αντλήσουμε διδάγματα και να βγάλουμε συμπεράσματα πολύ γρήγορα να σας μιλήσω για τη διαδικασία, γιατί νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν και τα επόμενα βήματα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας και με όλους. Μέχρι τα τέλη Νοέμβρη και λίγο το Δεκέμβρη έχω προβλέψει εγώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία των επαφών. Θα δούμε και αύριο τι, έχει, ε, τι έχουν να μας πει τα κράτη-μέλη και θα κάνουμε αξιολόγηση με βάση τα σχόλια που θα έχουμε λάβει μέχρι τότε για να δούμε για το τι μέλη γενέστε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Και υπάρχει λόγος για τον οποίο προβάλλονται αυτές οι δύο επιλογές. Προβάλλονται δύο επιλογές γιατί εκφράζουν διαφορετικές φιλοσοφίες. Οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές, θεμελιωτώς διαφορετικές και όταν μπει κανεί στις λεπτομέρειες η κατάσταση γίνεται πολύ πιο περίπλοκη. Δεν είναι το θέμα ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει πρόστιμο στο χύψη στη Γουατεμάλα και έτσι να αλλάξει το σύστημα. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό του κατά πόσο οι κυρώσει μπορούν πραγματικά να επιφέρουν αλλαγές στο εργασιακό ή περιβαλλοντικό περιβάλλον. Και έχουμε την ευθύνη να κάνουμε το σωστό. Γιατί σε τρία χρόνια πρέπει να μπορούμε να δείξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να φέρουμε την αλλαγή. Και το χειρότερο θα ήταν να σχεδιάσουμε ένα κακό μηχανισμό που τελικά να μην δουλεύει. Όλα αυτά ε, θα έχουν αντίκτυπο και στο πεδίο εφαρμογής. Μπορούμε να ονειρευτούμε και να κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια, όμως όλα αυτά επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής. Το Βιετνάμ δέχτηκε ένα πολύ μικρότερο πεδίο εφαρμογής δεσμεύσεων, ενώ με τις Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε ένα πολύ πιο ευρύ πεδίο δεσμεύσεων και αυτά θα εξαρτηθούν και από τους εταίρους που παρακολουθούν τη συζήτηση. Σε κάθε εμπορική συμφωνία έχουμε τη δοκιμή για τον αντίκτυπο στο εμπόριο. Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση της Γουατεμάλας και είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περάσει κανείς αυτό το τεστ όταν μιλάει για το περιβάλλον ή για τα εργασιακά. Πώς μπορεί να αποδείξει, ας πούμε, ότι η απουσία ελευθερίας, ελευθερίας του συνέρχεστε αποτελεί πλήγμα για το εμπόριο αυτό καθεαυτό. Τίθενται πολλά ερωτηματικά λοιπόν. Δεν λέω βέβαια ότι θα παρατήσουμε τελείως το ενδεχόμενο των κυρώσεων. Όμως, πολλές ε, από τις κοινότητες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τα εργασιακά ανησυχούν η ενεργή συμμετοχή είναι καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε τα ζητήματα, να τους εμπλέξουμε δηλαδή τους εταίρους μας. Π.χ. το κλίμα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πήγαν όλοι στο Παρίσι και συμφώνησαν εθελοντικά πάνω σε ένα σύστημα και αυτό το συμπεριέλαβαν, συμπεριέλαβαν στο FTA και το καθεξής. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν του Παρισιού ε, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει ε, αυτά τα συμφωνηθέντα, ειδικότερα από τη στιγμή που είπα αποσύρθηκαν από την ε, συμφωνία αυτή για το κλίμα. Αυτό που είναι απολύτως σαφές είναι ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Αυτό όλοι μας το λένε σε όλες τις ε, συζητήσεις μας. Όχι, δεν το αντιμετωπίζουμε καθόλου σαν να μην τρέχει τίποτα και δεν κάνουμε καθόλου business as usual. στο έγγραφό μας ε, έχουμε βάλει το feedback, την αντροφοδότηση από την οικονομική και κοινωνική κοινότητα, τους πολύ πεπειραμένους συμβούλους της ομάδες συμβουλευτικής, όλους που έχουν συντάξει έγγραφα για το πώς μπορούμε να εμπλέξουμε καλύτερα την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει στο έγγραφό μας, στο non-paper. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται προσφυγές. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Μεγάλο θέμα το θέμα του operation, της λειτουργίας, να μπορούν οι ομάδες συμβουλευτικής να λειτουργήσουν εντός των κοινωνιών, εντός των κρατών. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για διαφάνεια, αλλά υπάρχει και το θέμα της οικονομικής στήριξης. Μπορούν να συμμετέχουν αυτές οι ομάδες, να διαμορφώσουν, να επηρεάσουν την ατζέντα και ούτω καθεξής. Άπαξ και έχουμε λοιπόν ένα εργαλείο επίβλεψης ε, καλύτερα εξοπλισμένο, τότε θα μπορούμε εκ του σύνεκης να βλέπουμε κατά πόσο εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις. Σημειώνω και ένα άλλο παράπονο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ξεκίνησε μια διαδικασία επίλυσης διαφορά για, μια, για καμία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, για κανένα θέμα. Δεν έχουμε καμία εμπειρία πάνω σε αυτό. Κατανοώ όμως τα παράπονά σας και είμαι έτοιμη να πυροδοτήσω την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης διαφορών για την περίπτωση της Νότιας Κορέας. Οι διατάξεις είναι δεσμευτικές, αποτελούν και εκτιμένο, δεν έχουν ή εθελοντικό χαρακτήρα. Δεν ε, έχουμε αξιοποιήσει αυτό το μηχανισμό ε, με την Νότια Κορέα, αλλά είχαμε και αλλαγή κυβέρνηση και θέλησαμε να δώσουμε νέα ευκαιρία. Ευχαρίστως να το πράξουμε. Το ίδιο ισχύει και για την Ουατεμάλα Ενδεχομένω αυτή η περίπτωση που αναφέρατε περιλαμβάνεται στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Όμω μπορεί να μην λειτουργήσει λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτό το μηχανισμό επίλυσης διαφορών και μιλούμε για μια εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη. Βλέπω ότι τα κράτη-μέλη και εμείς συνεργαζόμαστε καλύτερα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και αυτό είναι σημαντικό και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μας παρακολουθεί και βλέπει ποια επίπτωση έχει η παρέμβασή μας. Βλέπετε λοιπόν ότι Σε πολλούς τομείς πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και τους εξετάζουμε προσεκτικά. Τώρα, για τις παλιές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, δεν ξέρω αν κατάλαβα το ε, ερώτημά σας. Από ό,τι γνωρίζω, ε, τα κεφάλαια για το εμπόριο και την αηφόρο ανάπτυξη βρίσκονται παντού. Ελπίζουμε να επανακινήσουμε τις διαπραγματεύσεις σύντομα με τις χώρες της Μεσογείου είτε την Ισία είτε άλλη χώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντοτε υπάρχει κεφάλαιο εμπορίου αηφόρου ανάπτυξης. Μεξικό και Χιλή ε, γίνεται διαπραγμάτευση για τα αντίστοιχα κεφάλαια εκεί. Στρέφομαι και προς τον συνάδελφο γιατί νομίζω ότι υπάρχει και στην Νότιο Αφρική και στην Αφρική Καραϊβική ε, Ειρηνικός Νομίζω ότι παντού έχουμε συμπεριλάβει τέτοιου είδου κεφάλαια. Για τη Γουατεμάλα να πω ότι πρέπει αυτά να τα έχουμε υπόψη όταν κάνουμε την αξιολόγησή μας. Τρία χρόνια μόνο ισχύει αυτή η συμφωνία με τη Γουατεμάλα. Τουλάχιστον ένα χρόνο χρειάζεται ε, μια χώρα για να θεσπίσει τις επιτροπές της. Οι ομόλογοι μας δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και εμπλοκή της στην ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Έχουμε άμεση επικοινωνία με συνομιλητέ. Τρία χρόνια χρειάστηκε η Γοτεμάλα να θεσπίσει το πλαίσιο για να μπορέσει να εφαρμόσει τη συμφωνία. Α του δώσουμε την ευκαιρία να το κάνουν. Προσωπικά είχα πάει μαζί με τον κύριο Λάγκε στο Βιετνάμ και εκεί πήραμε το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε ένα νωρίτερο στάδιο της διαδικασίας. Έχουμε εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο για να αυξήσουμε την πίεσή μας, την επιρροή μας πριν αρχίσει να ισχύει η Συμφωνία Ελευθερομπορίου για να μπει σε σωστές βάσεις και να δρομολογηθεί σωστά. Και όντω πρέπει να δράσουμε καλύτερα προληπτικά εκ των προτέρων. Ένα τελευταίο ερώτημα, μάλλον δεν το απάντησα, αλλά ξέρω ότι δεν έχετε και πολύ χρόνο. Με χαρά θα επανέλθουμε για να ξανασυζητήσουμε όλα τα ερωτήματα που θέτετε, τα ίδια ή και διαφορετικά. Να σας πω ότι είναι πολύ, πολλές και διαφορετικές οι απόψεις για το ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να επαναλάβω μια ερώτηση. Αναφέρατε τη βελτίωση ε, που βλέπετε στο non-paper και πέραν του ζητήματος της επιβολής και όλα αυτά φυσικά υπάρχουν κάποια βήματα βελτίωσης εκεί μέσα και υπάρχει και βελτίωση στο κεφάλαιο της στην ε, ΣΥΤΑ και το ερώτημά μου είναι πώς γίνεται τώρα η Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό να ε, προβάλλει ένα παλιό μοντέλο χωρίς τις βελτιώσεις αυτές. Δεδομένη τη κατάσταση που υπήρξε μέσα στο Κοινοβούλιο, ότι ήταν δύσκολο να επιτευχθεί πλειοψηφία ακόμη και για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Αν εγώ ήμουν η Κομισιόν, στη διαπραγμάτευση αυτή, θα έβαζα ε, αν μη τι άλλο, την επιτευχθήσα βελτίωση στο κεφάλαιο TST, διότι θα μπορούσε αυτό, να αποτελέσει, αυτό θα αποτελεί τη βάση για την ε, ε, διαπραγμάτευση και δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να έχει ως έκβαση κάτι χειρότερο από την αρχική μου πρόταση υπάρχει κίνδυνος να μην επιτύχω και πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί λοιπόν η Κομισιόν προτείνει στο Μεξικό και στις χώρες Μερκοσούρ τα παλιά έγγραφα που προέρχονται από συζητήσεις που έλαβαν χώρα πριν απο 3 3-4 χρόνια. Η δική μου αξιολόγηση είναι λίγο διαφορετική. Ε, υπό την εξή έννοια ότι στη ΣΥΤΑ και ξέχασα να απαντήσω την ερώτησή σας, ζητώ συγγνώμη για αυτό. Η ΣΥΤΑ πράγματι έχει τεθεί σε ισχύ. Προετοιμαζόμαστε για την ε, πρώτη ε, ανασκόπηση Πρέπει να βρούμε τις ημερομηνίε ουσιαστικά κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί, να δούμε και τα τεχνικά θέματα. Ο Καναδά είναι απασχολημένο με την αναθεώρηση τη ναύτα. Αυτή τη στιγμή απασχολεί όλε τι ομάδε. Η Κομισιόν επίση έχει γράψει και μια γενικού περιεχομένου επιστολή στον κύριο Σαμπάνη για να. και σκοπεύει να γράψει και μια επιστολή για την αναθεώρηση, για την ανασκόπηση το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε με τον Καναδά είναι να κάνουμε την ίδια συζήτηση αυτή, μαζί του, αυτή που κάνουμε εδώ τώρα. Ετίθεται και ένα ζήτημα χρόνου, διότι γίνεται μια συζήτηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ξέρω ότι εσεί έχετε τι δικέ σα απόψει, τι άκουσα προσεκτικέ, αλλά είναι πολλέ και διάφορε οι απόψει. Δεν μπορώ να πω ότι ε, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, ότι έχει καταλήξει κάπου. Είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί μέχρι του χρόνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωράνε τα πράγματα. Ε, και έχουμε και μια εξελισσόμενη ατζέντα. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Θα βάλουμε και ρήτρε αναθεώρηση με το Μεξικό και με τι Μερκοσούρ που θα τι έχουμε εμπνευστεί από τη ΣΥΤΑ ουσιαστικά. Ε, και αυτό προγραμματισμό να κάνουμε. Ε, όσον αφορά το κείμενο, είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς όλο. Αυτό που προτείνουμε, αυτές οι βελτιώσεις, είναι πράγματα που δεν χρειάζεται να αποτυπώνται στην ίδια συμφωνία. Όταν λέω ας πούμε θα δώσει τη δυνατότητα σε εσωτερικές συμβουλευτικές ε, ομάδες να δουλέψουν ε, Υπάρχει ένα ποσό τώρα 6 εκατομμυρίων ε, συμβόλων που θα ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτών των ομάδων. Αυτό δεν το συμπεριλαμβάνω μέσα στην συμφωνία. Πολλά πράγματα πρέπει να αποτυπώνται στα έγγραφα, σε διάφορα έγγραφα για να είναι ορατά, αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχουν και στις συμφωνίες. Ε, υπάρχει κάποιο προβληματισμό και εξακολουθούμε να λαμβάνουμε σχόλια με διάφορε ιδέε για το πώ θα εξορθολογήσουμε τα σχόλια που λαμβάνουμε από την κοινωνία των πολιτών πέραν τη εγχώρια συμβουλευτική ομάδα, πέραν των ενστάσεων κτλ. Το εξετάζουμε. Δεν έχω ακόμα απάντηση, αλλά δεν είναι κάτι που απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται στη συμφωνία. Σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να υποβάλει μια καταγγελία και των δύο εβδομάδων ε, ουσιαστικά, σε, σε, μόλις έλαβα και μια καταγγελία από μια ΜΚΟ για το Περού, για παράδειγμα. Όταν μιλάμε για τις βελτιώσεις του ΑΕΛΟ, δεν χρειάζεται αυτό να αναφέρεται συμφωνία, απλά πρέπει να φτιάξουμε μια διαδικασία σε αυτή την περίπτωση. Αυτή ίσως είναι η εξήγηση που χρειάζεστε. Και για το Παρίσι συζητήσαμε με τους Γάλλους, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, προτεραιότητα και για τον κύριο Μακρόν και ρωτάμε δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα κεφάλαια για το κλίμα και εμείς προτείναμε το εξή. είπαμε έχουμε θεσπίσει την αρχή στη συμφωνία και μετά χρειαζόμαστε ένα σχέδιο υλοποίησης που θα μας λέει τι ακριβώς θα κάνουμε για να βελτιώσουμε την κλιματική κατάσταση αυτό ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε δεν είναι παλαιομοδίτικη συμφωνία όπως τη λέτε, την επικαιροποιούμε απλά ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε τις συμφωνίες μας είναι ότι τις συμφωνίες μας θεσπίζουμε τις αρχές δεν εξηγούμε αναλυτικά όλες λεπτομέρειες Πρόεδρος, ναι, φυσικά. Ναι, αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Αλλά εάν συγκρίνω τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τη συμφωνία του Μεξικού, στη ΣΕΤΑ, για παράδειγμα, μία απέτηση ήταν να βελτιωθεί η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των βασικών προδιαγραφών του ILO και να δοθεί στους εργαζόμενους η δυνατότητα να προσφύγουν εάν παραβιάζονται οι βασικές, ε, τα βασικά τους εργασιακά δικαιώματα. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση στο Μεξικό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ε, μια τέτοια διάταξη για το Μεξικό. Γιατί δεν το προτείνει αυτό η Κομισιόν, εφόσον υπάρχει στη ΣΥΤΑ, γιατί δεν προτείνει κάτι παρόμοιο. Μπορείτε παρακαλώ να μου δώσετε μια απάντηση. Η Επιτροπή. Νομίζω ότι υποβλήθηκε μία λεπτομερής ερώτηση από τη Μόσκα μαζί με άλλες ερωτήσεις για τη ΣΕΤΑ θα μπορούσαμε να σας ξαναστείλουμε αυτές τις απαντήσεις. Και φυσικά θα σας στείλω και άλλες απαντήσεις για τις υπόλοιπες για να το διευκρινίσουμε. Δεν νομίζω ότι η κατάσταση για το Μεξικό είναι η υπολείπεται της κατάστασης ε, στη ΣΕΤΑ. Ευχαριστώ Μαντλέν, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι πεπισμένος ότι θα επανέλθουμε από αυτό. Και οι συντονιστέ αποφάσισαν να υπάρξει μια προφορική ερώτηση με ψήφισμα. Θα κάνουμε λοιπόν περαιτέρω βήματα για να εφαρμόζεται καλύτερα το TSD. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της σας διάταξης, το 23. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για την εφαρμογή της ε, διμερούς ρήτρας διαφύλαξης για τις μπανάνες. Ο κύριος Μάρτιν από το DigiTrade θα μας μιλήσει για τη διαδικασία εφαρμογής. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μας δίνει τη δυνατότητα να σας εξηγήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίηση για τι μπανάνε που περιέχεται στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Κολομβία, Περού, Εκουαδόρ και, και άλλων χωρών τη Κεντρική Αμερική ο μηχανισμός σταθεροποίησης γενικά λειτουργεί καλά. Μέχρι στιγμής είναι αποτελεσματικός. Οι τροπολογίες σε αυτό τον μηχανισμό που εισήχθησαν φέτος τη αιτήση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν εντάχθηκε και το Εκουαδόρ σε αυτή τη συμφωνία βελτίωσαν τη λειτουργία της συμφωνίας αυτής ούτω ώστε να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αν οι εισαγωγές φτάσουν στο 80% του ετήσιου ορίου τους. Και συχνά σας στέλνουμε στοιχεία για αυτές τις εισαγωγές με πιο εύχρηστη μορφή από τον προηγούμενο Απρίλιο. Η Γενική Διεύθυνση δημοσιεύει στον ιστοχώρο της κάθε εβδομάδα αναλυτικές πληροφορίες και πάλι εύληπτες. Η DigiTax επίσης έχει βελτιώσει την πρόσφαση τα στοιχεία για τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού σταθεροποίησης για τι μπανάνες. Σε καθημερινή βάση ενημερώνουν τα στοιχεία για τα πρόσφατα γεγονότα των εισαγωγές από την Ικαράγουα και την Γουατεμάλα. Υπερέβησαν αυτό το όριο το 80%. Το η συγγνώμη, η Επιτροπή τότε ενημέρωσε το Κοινοβούλιο το Συμβούλιο και την Αρμόδια Επιτροπή του στείλαμε τα τελευταία στοιχεία. Όταν φτάσαμε στο όριο του 100% η Κομισιόν έκανε μια μελέτη εμπεριστατωμένη για τις επιπτώσεις αυτών των εισαγωγών. Ιδιαίτερα εξετάσαμε εάν αυτές οι εισαγωγές ε, προκάλεσαν στρεβλώσεις στην αγορά ε, νοπής μπανάνας και καταλήξαμε <clears throat> ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια στρέβλωση και γι' αυτό η ο πρωτομησιακός δασμός των 97 ευρώ ανατόνου ε, που είναι πολύ μικρότερος από το δασμό των 222 ανατόνων που είναι ο δασμός του ΠΟΕ διατηρήθηκε. Το γεγονός ότι δεν ανεστάλλει λοιπόν αυτός ο πρωτομησιακός δασμός αποδεικνύει ότι λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός ο οποίος προβλέπει αυτή τη δυνατότητα δηλαδή αναστολής των πρωτομησιακών δασμών αλλά μόνο εάν υπάρξει κάποιος όγκος εισαγωγών. Αλλά δεν γίνεται αυτόματα, αιτιολογείται, εάν αυτές οι εισαγωγές μπορεί να προκαλέσουν σημαντική στρέβλωση στην αγορά. Γι' αυτό ο μηχανισμός καλεί την Επιτροπή να κάνει μια ανάλυση της επίπτωσης αυτών των εισαγωγών στην κατάσταση της ενωσιακής αγοράς για τις μπανάνες. Το γεγονό ότι ορισμένε τιμέ ε, ε, υπερβλήθησαν κατά τον ε, κατά την τρέχουσα κατά το τρέχον έτος μας αποδεικνύει ότι λειτουργεί το σύστημα προειδοποίησης για το τρέχον έτος το γεγονό ότι υπερβλήθησαν κατά λίγο τα όρια στην περίπτωση της Νικαράγουας και της Βατεμάλα ήταν 1,2% 1 έως 2% των συνολικών εισαγωγών Θεωρήσαμε λοιπόν ότι συνολικά δεν ε, δημιουργούνται στρεβλώσεις της ενωσιακής αγοράς. Αλλά στην περίπτωση της Νικαράγος που ήδη το Νοέμβριο φέτος σε σχέση με τον, ε, συγγνώμη, τον Μάιο φέτος, ενώ αντίθετα πέρυσι είχε υπερβεί αυτό το όριο μόλις τον Νοέμβριο, μόνο τον Νοέμβριο, Φέτος λοιπόν επειδή φτάσαμε στο όριο αυτό πολύ νωρίς, ε, κάναμε τις σχετικές προειδοποίησεις. Τώρα για το μέλλον αυτού του μηχανισμού σταθεροποίησης ο μηχανισμός λύγει στα τέλη του 19. Όμως υπάρχει δέσμευση στην κοινή διοργανική συμφωνία που λέει ότι η Κομισιόν θα εξετάσει την κατάσταση των παραγών μπανάνας πριν λήξει η ισχύση αυτού του μηχανισμού. Ιδιαίτερα θα εξετάσουμε εάν χρειάζεται επέκταση της περίοδου ισχύω. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα εξετάσουμε βέβαια και πώς θα διατηρηθεί η παραγωγή μπανάνας στην Ένωση, ιδιαίτερα στις ε, ιδιαίτερα απόμακρες περιοχές που υποφέρουν από ιδιαίτερα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στους εισηγητές. Ο κύριος Βίνκλερ θα αντικαταστήσει τον κύριο Μάτο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας διαβάσω την παρέμβαση του συναδέλφου Καμπριελ Μάτο για το ζήτημα αυτό. Το περασμένο Αύγουστο η Γουατεμάλα υπερεύει το κατόφλι που έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες. Η Νικαράγουα Επίσης το ξεπέρασε κατά 235%, το περί τρία χρόνια το ξεπερνάει, η Παναμάς, Κωνσταντίνα ξεπερνάνε το, το κατόφλι επίσης, το υπερβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλύσει την κατάσταση της αγοράς της μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της κατάστασης των παραγωγών πριν πυροδοτήσει το μηχανισμό αυτό Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν υπονομεύθηκε σοβαρά η κατάσταση των παραγωγών ούτε υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα της αγοράς. Όλα αυτά τεκμηριώνονται. Όταν δεν υπάρχουν νομικές επιπτώσεις αρνητικές δεν υπάρχει και αρνητική νομική δράση. Υπάρχει όμως πολιτική ευθύνη ενδεχομένως παρόλο που οι χώρες επανειλημμένως και προκλητικά ξεπέρασαν τα ε, κατόφλια, ως πολιτικός δυσκολεύομαι να δικαιολογήσω γιατί δεν αναλάβαμε δράση. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι οι παραχωρήσεις αυτές που δίδονται για τις μπανάνες είναι πέρα από τις παραχωρήσεις που ήδη δίνουμε στο επίπεδο του ΠΟΕ και έχουμε ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμό σταθεροποίησης και ούτε αυτά έχουν πυροδοτηθεί ποτέ, δεν έχουν αρχίσει να ενεργοποιηθούν και να ισχύουν. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε τους μηχανισμούς που συμφωνήσαμε και για διάφορους λόγους και για τον εξή λόγο. Αν δεν το κάνουμε, οι εξαγωγείς μπανάνες θα αξιοποιήσουν την αδράνειά μας και θα συνεχίσουν να εξάγουν παρά ε, και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν οι εξαγωγές αυξάνονται ασύστολα, ε, τότε αλλοιώνεται η ροή Ευχαριστούμε την Επίτροπο Μάλστρομ για τη δέσμευσή της και την ενεργητική της συμμετοχή για να ε, γίνει λειτουργικός ο μηχανισμός αυτός στο σημερινό. Υπάρχουν εναλλακτικέ όμως για το μέλλον. Ποιες είναι οι προτάσεις που έχει η Επιτροπή για το μέλλον ως εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και για τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της, για το τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί το μηχανισμό σταθεροποίησης ε, της αγοράς της μπανάνας, της εξόχως από κέντρες περιφέρειες. Ε, το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι Κανάριες νήσους εξαρτώνται τρόπον την υπερβολικά από την μπανάνα και εμείς είμαστε το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής στις Κανάριες νήσους. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε το θέμα στενά. Να πω ότι έχει βελτιωθεί πολύ η ροή των πληροφοριών μέσα από τα δελτία τα ενημερωτικά που δημοσιεύεται ως Επιτροπή στον τοπό σα. Θέλω όμως να σας ζητήσω καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει απλά να μας δίδετε τα στοιχεία για τους παραγωγούς και αντίστροφα, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αν δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία δίδετε εσείς μόνο στους παραγωγούς. Πρέπει να, με πιο συχνό τρόπο και με πιο πολλές λεπτομέρειες να είμαστε το, αυτό που με ανησυχεί είναι το εξή. Στη συμφωνία με την Κεντρική Αμερική ε, προοδευτικά μειώνονται οι δασμοί που θα ισχύσουν για την μπανάνα και θα ξαναμειωθούν στα 75 ευρώ τον τόνο από την 1η Πρώτου του 2020. Ο μηχανισμός σταθεροποίησης λύγει στα τέλη του 2019. Άρα θα είχαμε την, το 2020 την εξή κατάσταση. Θα μειωθεί μόνιμα, μόνιμη μείωση των δασμών και απουσία μηχανισμού σταθεροποίησης. Είναι λογικό, ε, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια αξιολόγηση από πριν. Εξάντε, πάντοτε πρέπει να αξιολογείται όλο κάθε σύστημα λειτουργίας, όμως έχουν χτυπήσει τα, καμπανάκια του συναγερμού, ε, στην Ικαράγου ας πούμε, φάνηκε ε, το Μάιο ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο μηχανισμός. Δεν είναι δυνατόν ένας κλάδος τόσο ευάλωτος να μην είστε βέβαιοι ότι ο μηχανισμός θα δουλέψει πάντοτε. Ιδαλλιώς θα έχουμε πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις εξόχως απόκεντρες περιφερειές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Κανάριες νήσους, νήσι, όπου οι οικογένειες ολόκληρες εξαρτώνται. Ε, η οικονομική του δραστηριότητα εξαρτάται από την μπανάνα. Οι τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κατόφλια για ε, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης λειτουργήσαν, ήταν πολύ χρήσιμες και αποδείχθηκε η χρησιμότητά τους. Σας ζητώ λοιπόν να μας ακούτε με περισσότερη, με μεγαλύτερη προσοχή γιατί όταν προτείνουμε κάτι ε, έχουμε ειδικό βάρος και το προτείνουμε για κάποιο λόγο πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτσπαρκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την ενημέρωση και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε έγκαιρα αυτές τις ε, προειδοποίησεις, τις έγκαιρες προειδοποίησεις για να μπορούμε να αντιδράσουμε. Όμως, ορισμένοι θέτουν ε, το θέμα της εξάρτησης της παραγωγής μπανάνας. Και τώρα θα σας πω κάτι το οποίο θα σας φανεί τολμηρό. Καλούμε τις τρίτες χώρες ε, να αναπτύξουν νέε μεθόδου προϊόντων, να ε, καλλιεργήσουν άλλα προϊόντα για να είναι αυτόνομοι. Τι κάνουμε εμεί όμω για με τη δική μα παραγωγή μπανάνα σε αυτέ τι ε, εξόχω απόμακρε περιοχέ. Πρέπει να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Τι προοπτικές δίνουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε για τις μπανάνες του ε, fair trade δικαίου εμπορίου και για τις ε, βιολογικές μπανάνες. Πώς μπορούμε λοιπόν ε, να βοηθήσουμε την παραγωγή μπανάνας να αποκτήσει προστιθέμενη αξία. Και θα συμπεριλάβουμε βέβαια και το θέμα της ρήτρας διαφύλαξης. Άρα δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο η ποσότητα της παραγόμενης μπανάνας αλλά πρέπει να γίνει μία και ποιοτική βελτίωση. Να θέσουμε νέες προδιαγραφές. Να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής, αλλά και κατανάλωση της μπανάνας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν περαιτέρω επιχειρήματα. Πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από το υπάρχον σύστημα. Να κάνουμε νέες προτάσεις. Πρέπει να αποτιμήσουμε. ούτως ώστε να υπάρξει αυτόνομη ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ανταλλάξαμε λοιπόν απόψεις και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της μπανάνας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Το αγαπημένο μου θέμα σε κάθε ημερήσια διάταξη είναι τα διάφορα. Δεν υπάρχει κανένα. Και το τελευταίο. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου. Θα τα πούμε τότε.